Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ που ήρθατε στη συνεδρίαση της Επιτροπής μας, Εγκέρος. Αρχίζουμε αμέσως. Όσοι είστε, επιτρέψτε μου να ανακοινώσω ότι αναμεταδίδεται στο διαδίκτυο η συνεδρίασή μας ε, και για τη διερμηνία δίνεται προτεραιότητα στις γλώσσες των τακτικών μελών της Επιτροπής ε, υπο, ε, ΣΕΝΤΕ, Υποεπιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας. Εγκρίνουμε την μίληση διάταξη αν δεν έχετε αντιρρήσει σχόλια. Ωραία, εγκρίθηκε. Ανακοινώσεις της Πρόεδρου. Uh, Will have, unfortunately. <coughs> Δυστυχώς, ο πρέσβης, ο κύριος Σεράνο, πρώτος ομιλητής, θα πρέπει να φύγει στις 10 παρατέταρτο ακριβώς λόγω άλλων ανηλυμένων ε, υποχρεώσεων. Οπότε οι ερωτήσεις και απαντήσεις θα είναι πιο σύντομες. Ε, θα κάνουμε λοιπόν ένα διάλειμμα ενός τετάρτου 10 παρατέταρτο με 10 για να αρχίσει στις 10 η κοινή ακρόαση με την Επιτροπή Εξωτερικών και διάφορες αντιπροσωπείες που έχουμε ε, με την περιφερειακή. Γνωρίζετε ότι η ακρόαση αφορά τη Βόρεια Κορέα. Άλλη ανακοίνωση. Στο Στρασβούργο στις 14 ε, Δεκεμβρίου θα έχουμε μια ειδική έκτακτη συνεδρίαση για να συζητήσουμε τις τροπολογίες για την ομοδότηση του κυρίου Πάσκου. Ωραία. Ε, ευχαριστώ. Χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση θέλω να δώσω το λόγο στον πρώτο μας ομιλητή, ο οποίος είναι απριωτής γενικός γραμματέας ε, της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, ΕΙΕΔ, είναι ο πρέσβης κύριος Πέντρο Σεράνο, ο οποίος θα μας ενημερώσει ε, για ε, τις συζητήσει και τα αποτελέσματα ε, του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της 13 η Νοεμβρίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη που είναι τόσο ε, τσιμωγμένο το πρόγραμμά μου και στεναχωριέμαι και εγώ γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το πρωινό. Ε, το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων του Νοεμβρίου, όπως γνωρίζετε, ήταν μια σημαντική στιγμή για να προχωρήσουμε την, ε, το θεματολόγιο της άμυνας. Είναι κάτι το οποίο θα επιβεβαιωθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θα ήθελα όμως να σας ενημερώσω για το πώς ε, ε, πηγαίνουν τα πράγματα. Στις 13 Νοεμβρίου ασχοληθήκαμε με τρία βασικά στοιχεία. Πρώτο πρώτο ήταν εκτός του επίσημου συμβουλίου που ήταν ε, η υπογραφή από 23 κράτη-μέλη, οι περισσότεροι ήταν Υπουργοί ε, Αμήνης και Εξωτερικών, για την πρόθεση συμμετοχή μιας ε, μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας στον τομέα της άμυνας Υπέγραψαν λοιπόν μια κοινοποίηση και εξέφρασαν την θέλησή τους να προχωρήσουν ε, σε σχέση με το θέμα αυτό και κατά πάσα πιθανότητα τη Δευτέρα, την στο επόμενο ε, Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, ε, η ΠΕΣΚΟ, αυτή η μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία, θα εγκριθεί. Το κείμενο το οποίο υπεγράφει στις 13 Νοεμβρίου ε, περιέχει κάποιες αρχές όσον αφορά τη συνεργασία και ένα πρώτο σύνολο ιδεών σε σχέση με την ε, διαχείριση αυτής της ε, συνεργασίας. Μετά την υπογραφή αυτή ε, έγινε μια συνεδρίαση Υπουργών ε, Άμυνας και Εξωτερικών σε μεσημεριανό γεύμα και ήταν μια ευκαιρία να εξεταστούν όλες ε, οι πτυχές αυτές, αυτής της συνεργασίας. Επικεντρώθηκαν περισσότερο στην άμυνα, στην συνεργασία, την ανάπτυξη των αμυντικών ικανοτήτων. Όπως γνωρίζετε η ΠΕΣΚΟ, η μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία, αυτό αφορά. Συζητήθηκαν, συζητήθηκαν επίσης θέματα για τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Αμυντικού Αμυντικού Ταμείου που θα φτάσει και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύντομα φαντάζομαι. Εν πάση περιπτώσει πρέπει να υπάρχει μια συμφωνία και γι' αυτό σε κάποια μορφή. Όσον αφορά τώρα το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ε, Άμυνας ε, και αμυντικής ε, βιομηχανίας. Είναι, πρόκειται για στοιχεία που πρέπει να λειτουργήσουν από, από κοινού. Είναι κάτι το οποίο ε, τονίστηκε στα συμπεράσματα του Εξωτερικού Συμβουλίου ε, και είναι κάτι το οποίο θα ξανασυζητηθεί. Είναι πάρα πολύ σαφές αυτό γιατί η μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία θα συμπεριλάβει προγράμματα ανάπτυξης αμυντικών ικανοτήτων και είναι σημαντικό να μπορούν να είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση μέσω του Ευρωπαϊκού Αμυντικού Ταμείου και η αιτήσια αναθεώ θα βοηθήσει να εντοπίσουμε κενά στην ε, αμυντική ικανότητα του, στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Αμυντική Ικανότητα και την ανάπτυξή του. Όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν συνδέονται μεταξύ τους ε, πολύ στενά. Μετά ε, το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ε, άρχισαν να δημιουργούνται κάποιες γέφυρες για να υπάρξει μια ε, συνεργασία μεταξύ της ΠΕΣΚΟ αλλά και των οργάνων χρηματοδότησης με ιδιαίτερη βαρύτητα στην συνεργασία, κάτι το οποίο τόνισε και ύπατη εκπρόσωπος μεταξύ των διαφόρων πρωτοβουλειών και όπως γνωρίζετε επίσης οι δομές ε, της μόνιμης ε, διαρθρωμένης συνεργασίας βασίζονται σε ομάδες εργασίας του Συμβουλίου, σε σύνθεση ΠΕΣΚΟ, e που σημαίνει βέβαια ότι όλοι όσοι συμμετέχουν σε αυτές τις ε, ομάδες εργασίας θα συμμετέχουν και στις ομάδες εργασίας της ΠΕΣΚΟ. E Τη Δευτέρα, που μας έρχεται. Δεν περιμένουμε μόνο την έγκριση της επίσημης απόφασης για τη δημιουργία της ΠΕΣΚΟ, αλλά και την ανακοίνωση των πρώτων προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν μέσω της ΠΕΣΚΟ και αυτό θα είναι κατά πάσα πιθανότητα δήλωση ε, στα κράτη που συμμετέχουν στην ΠΕΣΚΟ 18 ε, projects έχουν ε, ε, θεωρηθεί μια πρώτη ομάδα προγραμμάτων που θα εξεταστούν. Θέλουμε να μην μείνουμε μόνο στις, διαπραγμα... διαδικασίες και στην γραφειοκρατία. Θέλουμε να γίνει πραγματικότητα και να υπάρξει μια πραγματική αμυντική ικανότητα που θα προκύψει από τη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία. Άλλοι τομείς ε, που συζητήθηκαν ε, της ε, εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας ήταν ας πούμε η πολιτική πλευρά. Όπως ξέρετε αυτό έχει γίνει πάρα πολλές φορές, έχει, πει, έχει υπάρξει πίεση και από διάφορες επίγουσες καταστάσεις το είδαμε δηλαδή από την αρχή ότι η ΕΠΑ η πολιτική ε, αφορά τα δύο τρίτα των ε, αποστολών μας, οι οποίες είναι πολιτικού χαρακτήρα και όχι στρατιωτικού χαρακτήρα και παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην, στην μεταρρύθμιση κάποιων τομέων, όπως για παράδειγμα στο Κωσυφοπαίδιο. Κάποια κράτη-μέλη θέλουν λοιπόν να εξετάσουμε εις βάθος το πολιτικό αυτό κομμάτι της ΕΠΑ για να δούμε πώς προσαρμόζεται καλύτερα στην αντιτρομοκρατία, ε, στον υβριδικό πόλεμο, στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος ή ε, του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο. Είναι δουλειά που έχουμε ήδη ε, δρομολογήσει. Η ανάπτυξη των ικανοτήτων πολιτικού χαρακτήρα είναι διαφορετικές από τις αμυντικές ικανότητες. Συνήθως στις αμυντικές ικανότητες μιλάμε για υλικό ε, στο, πολιτικό κομμάτι είναι πολύ σημαντικός ο ανθρώπινος παράγοντας και η μεγαλύτερη πρόκληση ε, είναι ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν σε όλα τα κράτη-μέλη για ε, εσωτερική χρήση και όχι τόσο για προβολή προς τα έξω. Ε, η περίοδος τώρα των, ε, του οικονομικών περιορισμών είναι ε, τέτοια που είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτρέπει να υπάρχουν υπεράριθμοι δικαστές, αστυνο, αστυνομικοί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο λοιπόν να αποσταλούν δικαστές ή αστυνομικοί εκτός των συνόρων για τέτοιου είδους αποστολές και αυτό είναι κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Αυτό που κάνουμε τώρα είναι να υπάρχει ένα έγγραφο αρχικό που θα ορίζει ε, τους στόχους και τις ε, αρχές του πολιτικού ε, τμήματος της ΕΠΑ και επίσης πρέπει να έχουμε και ένα πρόγραμμα ανάπτυξης που θα καλύπτει το πλήρες φάσμα όλων των αποστολών, αλλά κυρίως ε, τις βασικές προτεραιότητες που ανέφερα ήδη. Ο στόχος είναι, σε σχέση με τις εντολές που λάβαμε από το Συμβούλιο, είναι να οδηγηθούμε σε μια σε ένα σύμφωνο ε, πολιτικής ΕΠΑ ε, που ε, θα ορίζει όλα αυτά τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τις αποστολές αυτές. Και βέβαια πολύ σημαντικό είναι η σχέση μεταξύ των αποστολών ΕΠΑ και των νέων ρόλων πολιτικών αποστολών του ΕΠΑ που είναι εκτελεστικού ή με εκτελεστικού χαρακτήρα. Βλέπετε μερικέ φορέ ότι όταν πηγαίνουμε σε αυτέ τι πολιτικού χαρακτήρα αποστολέ που μπορεί να συμπεριλαμβάνουν για παράδειγμα έρευνε στο πλαίσιο μια ποινική διαδικασία. Ε, υπάρχει δηλαδή πάντοτε μια, σε μια συγκεκριμένη διάσταση ε, σε αυτέ τι αποστολέ που είναι μη εκτελεστικέ. Είναι ένα υβριδικό ε, μια υβριδική ε, πολιτική ΕΠΑ, ε, για να το πω έτσι. Αυτό είναι κάτι που θα ήθελα να τονίσω λοιπόν σήμερα. Άλλα πράγματα τα οποία συζητήθηκαν είναι πίεση για περισσότερη γενεοδορία στον καθορισμό του κοινού κόστους, στον μηχανισμό Αθηνά είναι κάτι το οποίο βέβαια στο οποίο έχουμε κάνει λίγη πρόοδο αλλά χρειάζεται περισσότερη ε, η στρατιωτική κινητικότητα είναι κάτι που επίσης είναι σημαντικό. Το συζητήσαμε στις, συζητήθηκε στις 13 Νοεμβρίου. Ε, η κινητικότητα εντός της Ευρώπης ε, και η ευθύνη των κρατών μελών βεβαίως. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ζητήσει αλλαγές διαδικασίες, στους κανονισμούς, στην ανάπτυξη των υποδομών που μπορούν να διευκολύνουν την κινητικότητα των δυνάμεων εντό τη Ευρώπη. και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το έχει ζητήσει και το ΝΑΤΟ. Είναι σημαντικό ε, επειδή αφορούσε και το δεύτερο τμήμα τη συνάντηση, που ήταν η συνεργασία Ευρωπαϊκή Ένωση ΝΑΤΟ. Έχει όμω και μια ευρωπαϊκή πλευρά. Η κυβερνοάμυνα επίση είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, η σχέση μεταξύ της κυβερνοασφάλειας και της άμυνας στον κυβερνοχώρο και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό κατά το ερχόμενο έτος είναι πέραν πάσης αμφιβολίας ότι αυτή η κυβερνοάμυνα είναι κάτι που θα μας απασχολήσει πολύ. Ε, όσον αφορά τώρα την ε, συνάντηση Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ, για τη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ, ε, Συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας, όπω γύφιστε πλέον. Πρέπει να σκεφτούμε λιγάκι με το βλέμμα στο μέλλον το Συμβούλιο ενέκρινε ένα νέο σύνολο κοινών προτάσεων ε, για τη συνεργασία με τον ΝΑΤΟ, 32 ε, αναδιάρθρωση τομέων που εντοπίστηκαν, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη στρατιωτική κινητικότητα, ε, στην αντιτρομοκρατία, και συνεργασία μεταξύ εταίρων για την καταπολέμηση της τροποκρατίας, ο κυβερνοχώρος, ε, η, ε, το 2018 η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια μεγάλη πρόκληση να αντιμετωπίσει γιατί θα έχει ηγετικό χαρακτήρα, ηγετικό ρόλο, ε, συγγνώμη, στην, στο συντονισμό των παράλληλων ασκήσεων. Σημαντικό σημείο ε, για το ΝΑΤΟ είναι πώς αυτές οι ικανότητες που αναπτύσσονται μέσω αυτών των νέων μέσων της ΠΕΣΚΟ, του Ταμείου για την Άμυνα, πώς θα είναι υποφελή όλα αυτά και για το ΝΑΤΟ, όχι μόνο ως προς τις δεσμεύσεις, μεταξύ των οποίων είναι η αύξηση, για παράδειγμα, της επένδυσης στον τομέα της άμυνας και μεγαλύτερη δέσμευση για την ανάπτυξη ε, ικανοτήτων αμυντικών. Ε, το ΝΑΤΟ ήταν λοιπόν πάρα πολύ θετικό. Προφανώ υπάρχει ένα σύνολο δυνάμεων, τα κράτη-μέλη έχουν ένα σύνολο δυνάμεων, ε, το οποίο σημαίνει ότι ό,τι του ωφελεί στο πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα του ωφελεί και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Αυτό είναι κάτι που αναγνωρίζει το ΝΑΤΟ και μάλιστα και την περασμένη Τρίτη στην συνάντηση των ε, Υπουργών ε, Εξωτερικών στο Συμβούλιο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας ε, την παρουσία των Υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών. Επίση, οι προδιαγραφέ που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, ώστε ό,τι και να γίνει στο πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, να ε, ωφελεί και την κινητικότητα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Ότι χρειάζεται, ό,τι γίνεται ήδη στο ΝΑΤΟ δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνεται και σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει υπάρξει λοιπόν πολύ σημαντική πρόοδο ω προ αυτό. Ε, όλα αυτά θα ξανασυζητηθούν στο Ευρωπαϊκό ε, Συμβούλιο το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Και νομίζω ότι θα τονιστεί ιδιαίτερα και η σημασία της εφαρμογής της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας και το θέμα της συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ. Αν δούμε, πούμε, το χρόνο που θα έχουμε μπροστά μας, ε, ε, η εφαρμογή είναι πάρα πολύ σημαντική. Έχουμε αναπτύξει πολλές πρωτοβουλίες, ο κανονισμός του EDIDP θεωρούμε ότι θα περάσει ομαλά και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ελπίζουμε εντός του πρώτου εξαμήνου και επίσης η συνοχή μεταξύ των εργασιών μας ε, και συνεργαζόμαστε μάλιστα και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις πολλές προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Η εφαρμογή λοιπόν και η συνοχή μεταξύ των δράσεών μας είναι νομίζω οι δύο βασικοί ε, όροι που θα περιγράψουν την επόμενη χρονιά. Επίσης, αύξηση του, ε, του, του ε, αποτελέσματος που επιφέρουμε επί τόπου. Έχουμε πάρα πολλές αποστολές. Θα υπάρξει λοιπόν Ειδικότερα στο Σαχέλ είναι πάρα πολύ σημαντικό το τι κάνουμε στο πλαίσιο της ΕΠΑ. Είναι σημαντικό να κινητοποιήσουμε όλα τα μέσα συνεργασίας που έχουμε στη διάθεσή μας, να σταθεροποιήσουμε μια περιοχή που είναι πάρα πολύ σημαντική για την Ευρώπη. Είναι πολύ σημαντικό κατά τη διάρκεια του 2018 για τις χώρες ε, του G5 και του ε, Σαχέλ είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και ε, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ οι διαπραγματεύσεις αυτών των κοινών προτάσεων είναι κάτι το πάρα πολύ περίπλοκο, μια πολύ περίπλοκη διπλωματική διαδικασία και έχουμε με πάνω από 74 τώρα ε, δράσεις έχουμε πάρα πολλά, ε, πολλές αποστολές ε, να περάσουμε μια πολύ πλούσια γεμάτη ζωή συνεργασίας με τον ΝΑΤΟ. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να συνεργαστούμε και εκεί θα επικεντρωθούμε κατά το επόμενο έτος. Με πολύ χαρά λοιπόν σας έκανα αυτή την παρουσίαση και ευχαρίστω αξιότιμοι ευρωβουλευτές να απαντήσω σε ερωτήσεις σας τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ξοχότατε. Πρέσβη κύριε Στεγάνο, σας ευχαριστώ για την ενημέρωση αυτή. σχετικά με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων με συμμετοχή των Υπουργών Εξωτερικών και των Υπουργών Μήνης, αργότερα με μέλη του ΝΑΤΟ. Σας ευχαριστώ για την τακτική και συχνή σας συμμετοχή εξ όσων ε, θυμόμαι είχατε έρθει και τον Ιούνιο. Πρώτος ο κύριος Γκάλερ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την αναφορά αυτή του πεπραγμένου συμβουλίου. Μια ερώτηση που θα πρέπει να ρωτήσω και τον Υπουργό ε, Ζούντα αμέσως μετά. Τι γίνεται με την ε, ενεργοποίηση της μόνιμης διαρθωμένης συνεργασίας και τη χρηματοδότησή της. Το άρθρο 41 θα εφαρμόσει το Συμβούλιο που λέει ότι τα διοικητικά ε, έξοδα και τα επιχειρησιακά εκτός από τις στρατιωτικές δαπάνες καλύπτονται από τον ε, προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το άρθρο θα χρησιμοποιηθεί. Ε, σας ενθαρρύνω πολύ να το χρησιμοποιήσετε αυτό γιατί αλλιώ θα χρειαστεί ομόφωνη απόφαση για να αποκλίνετε. Είναι πολύ σημαντικό για μας το Κοινοβούλιο και αν Τώρα δυστυχώς έχω στο γραφείο μου την Υπουργό να με περιμένει, θα πάρω να τη ρωτήσω τα ίδια και θα πάρω την απάντηση από τους συναδέλφους. Λυπάμαι πάρα πολύ. Okay. Ο κύριος Σδρογεύσκη τότε λοιπόν. E, tak, ja chciałem zadać pytanie kontynuujące pytanie kolegi Galera. Jak będą rozkładały się να συνεχίσω από την ερώτηση που έκανα κύριος ε, Γκάλε. Τι γίνεται με τον προπολογισμό αρχής δεδομένη από τις διοικητικές δαπάνες. Γιατί ακούμε και ποσά πολύ σημαντικά. Πώς θα ρυθμιστούν αυτά τα δημοσιονομικά θέματα. Η Πρόεδρος. Δεν ξέρω αν θέλει το λόγο ο κύριος Σαφοζέρ. Ε, παρακαλώ ζητήστε το αν θέλετε να πάρετε το λόγο, γιατί έχω και εγώ να κάνω κάποια ερώτηση. Στην περασμένη μας ε, ερώτηση, ε, συνάντηση, μάλλον μιλήσατε για τρεις τομείς πιλωτικής συνεργασίας για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Μολδαβία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη και την Ισία. Είναι τρει περιοχές και τρει χώρες με τις οποίες συνεργαζόμαστε με το ΝΑΤΟ για την ασφάλεια, την ηλεκτρονική και διαδικτυακή. Εκεί τι δράσεις αναλαμβάνονται και τι μπορείτε να μας απαντήσετε ως προς τα επιτεύγματα ή τα αποτελέσματα των δράσεων αυτών. Ποιος θέλει το λόγο. Α, κύριο Σαφοζέρ. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Γραμματέα και κυρία Πρόεδρε. Κύριε Γενικέ, ε, καθυστέρησα λίγο και ζητώ συγγνώμη. Ήθελα όμως να σας κάνω μια ερώτηση, η οποία μπορεί να μην είναι πάρα πολύ εύστοχη σκόπιμη σε σχέση με τα όσα είπατε. Αλλά ε, με ενδιέφερε να μάθω το Συμβούλιο. Πώς προβληματίζεται με τα νέα δεδομένα στις ΗΠΑ. Ο πρόεδρος Τραμπ μας καλεί να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και ζητεί να είμαστε ε, πραγματικοί, έτσι, γνήσιοι εταίροι. Αυτό κανονικά θα πρέπει να οδηγήσει στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ε, συστήματος. Γιατί όταν είσαι υπεργολάβος, εταίρος δεν νοείσαι. Και πρόσφατα διάβασα ένα βιβλίο πάρα πολύ ωραίο και το συνιστώ σε όλους, ο Αμερικανός φίλος του Μισελ Μπρανκάι, ο οποίος είναι ιστορικός και έλεγε ότι στη συνθήκη των Ηλυσίων για τη γαλλογερμανική ε, ενότητα 24 Ιανουαρίου 1963 το ΝΑΤΟ δεν συμπεριλαμβανόταν σε αυτή τη συμφωνία και μετά επίεσαν οι Αμερικανοί και ο Μονέ και ο κύριος Μονέ για να συμπεριληφθεί και το ΝΑΤΟ. Αρχικά όμως όταν βάζαμε τα θεμέλια για την Ευρώπη στο γαλλογερμανικό δίδυμο, ε, σκεφτόμασταν να δημιουργήσουμε μια Ευρώπη ανεξάρτητη του ΝΑΤΟ για την ασφάλεια και την άμυνά της. Ανεξάρτητη δεν σημαίνει ότι δεν ήμασταν εταίρος του ΝΑΤΟ. Ο στρατηγός Ντεγκόλ ήταν ο πρώτος ε, που παρενέβη και απουσίαζαν κάποιοι άλλοι. Και είναι σημαντικό να το γνωρίσουμε όταν ε, έγινε εισβολή στο Βερολίνο. Ήθελε να στείλει αμέσως τα γαλλικά άρματα αλλά από τους Άγγλους και τους Αμερικανούς δεν απαντούσε κανείς το τηλέφωνο. Αυτό νομίζω είναι το κλειδί για την ευρωπαϊκή επανίδρυση. Ευχαριστώ. Κύριε Πρέσβη, νομίζω πολλές ήταν οι ερωτήσεις και σας παρακαλούμε να απαντήσετε. I, do not δεν βλέπω να υπάρξει δεύτερος γύρος ερωτήσεων. Θα δούμε. Παρακαλώ, όσο χρόνο θέλετε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά το κόστος ε, της μόνιμης διαθρωμένης εργασίας της ΠΕΣΚΟ και τη λειτουργία της, κοιτάξτε, βασιζόμαστε στο εξή ότι πρέπει να μειώσουμε τις επιπρόσθετες διοικητικές δαπάνες, και επίση ε, πρέπει να αποφύγουμε να προκύψει νέα γραφειοκρατική επιβάρυνση. Δηλαδή, κατ' ουσίαν η ΠΕΣΚΟ ε, θα λειτουργήσει με ό,τι έχουμε στη διάθεσή μας. Βεβαίως, ε, ενδεχομένως να χρειαστεί κάποια ενίσχυση σε επίπεδο προσωπικού. Θα το δούμε λιγάκι αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι δεν θα υπάρξει μια ειδική υπηρεσία, ειδική μονάδα για την ΠΕΣΚΟ. Η υπηρεσία εξωτερική δράση, το στρατιωτικό προσωπικό προσωπικό ή ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας. Από εκεί θα εντοπιστούν, θα αποσπαστούν ίσως κάποιοι υπάλληλοι οι οποίοι θα υπηρετήσουν την ΠΕΣΚΟ. Και αυτοί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι ήδη ασχολούνται με την ανάπτυξη των αμυντικών ε, ικανοτήτων. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν θα υπάρξει πουντενή ουσιαστική αλλαγή. Θα έχουμε δηλαδή την φυσιολογική ενίσχυση μιας υπηρεσίας ε, η οποία θα αναλάβει κάποιες επιπρόσθετες αρμοδιότητες στο πλαίσιο της δουλειάς που έτσι κι κάνει. Αυτά όσον αφορά στο διοικητικό κόστος. Όσον αφορά το κυβερνοστοιχείο, εξετάζουμε το θέμα της ε, κοινής επικοινωνίας, το οποίο τέθη το Σεπτέμβρη και το οποίο έχει κάποια εξωτερική επίσης διάσταση, δηλαδή αγγίζει την ε, κυβερνόμηνα. Και επίσης, όπως πολύ σωστά είπατε, αυτό που εξετάζουμε είναι το πώς ε, μπορούμε να στηρίξουμε τους εταίρους μας για να αναπτύξουν τις δικές τους κυβερνοδυνατότητες. Στη Μόλδοβα, όπως ξέρετε, Μολδαβία μάλλον, εκεί έχουμε μια άσκηση όπου εξετάζεται η αντίσταση που μπορεί να υπάρξει σε αυτό το υβριδιακό πλαίσιο. Εκεί είναι μια χώρα που έχουμε κάνει μια πολύ σημαντική μελέτη και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε και με άλλους. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε, όπως ήδη το έχουμε πράξει, στο πλαίσιο της αντιτρομοκρατίας να έχουμε ένα κοινό πρόγραμμα πρόγραμμα Σε αυτά τα θέματα δουλεύουμε τώρα και βέβαια θα ε, συνεχίσουμε να δουλεύουμε διότι θεωρώ ότι για το θέμα αυτό μπορούν ε, να προκύψουν ακόμα πάρα πολλά στο επίπεδο των δυνατοτήτων. Με το τελευταίο σας ερώτημα για τη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ και πώς αναπτύσσουμε και την Ευρωπαϊκή Άμυνα. Σύμφωνα απολύτως. Δεν υπάρχει καμία αντίφαση. Έχει το ΝΑΤΟ ρόλο να διαδραματίσει τον οποίο δεν αφισβητεί κανείς αυτή τη στιγμή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χρειάζεται ίδια μέσα ασφάλειας και άμυνας. Είχε γίνει μια πολύ θεωρητική συζήτηση, όπως θα ξέρετε, φαντάζομαι, ε, στην αρχή του 2000. Αυτό που τότε ονομαζόταν Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας, ΕΠΑ, και υπήρξαν πολλοί φόβοι, όχι μόνο στο ΝΑΤΟ, αλλά και στον ΟΗΕ. Δηλαδή μήπω οι προσπάθειες που κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν εις βάρος ε, τη συμμετοχή μα στο ΝΑΤΟ και εις βάρος επίσης τη συνεισφορά των κρατών μελών ε, στο ΝΑΤΟ, στον ΟΗΕ στις ε, αποστολές. Αλλά όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν έδωσαν την απάντηση, η οποία απάντηση λέγει ότι πρώτον χρειαζόμαστε αυτές τις ευρωπαϊκές ικανότητες και Ε, οι ικανότητες αυτές έρχονται να καλύψουν κάποιες ελλείψεις και κάποια ελλείμματα ε, στην άμυνα και στην ασφάλεια που δεν μπορεί να καλύψει το ΝΑΤΟ από την ίδια του τη φύση και τις δομές του. Άρα κλείνουμε αυτό το κενό που υπάρχει από τη μια και από την άλλη. Αυτό φυσικά δεν είναι εις βάρος της συμμετοχής μας στο ΝΑΤΟ ή στον ΟΗΕ. Και μια πιο πρόσφατη εξέλιξη βλέπουμε τώρα πώς και πόσο μπορούν οι προσπάθειες που κάνουμε να βοηθήσουν στην ανάπτυξη ικανοτήτων. Εντάξει, τότε δημιουργήσαμε τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας και δεν ξέραμε πάρα πολύ καλά πώς θα λειτουργούσε, αλλά τώρα με τις νέες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται, Έχω την αίσθηση ότι το ΝΑΤΟ ποντάρει πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να ε, πιέσει και να προωθήσει την ανάπτυξη ικανοτήτων των κρατών μελών. Άρα τα κράτη-μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις δυνάμεις και στο ΝΑΤΟ και στον ΟΗΕ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το στοιχείο που προσθέθηκε τώρα πιο πρόσφατα, μετά το 2011 ας πούμε, και μετά όλες αυτές τις κρίσεις που γνωρίσαμε και που αδέξια χαρακτηρίσαμε ε, ε, Αραβική Άνοιξη, είδαμε ιδιαίτερα μετά το 2014 ότι, ότι χρειάζεται επιπλέον ε, ίδια ε, ε, ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχω την αίσθηση ότι το ΝΑΤΟ δεν το βλέπει αλλιώς γιατί τώρα βρισκόμαστε στην καλύτερη φάση των σχέσεών μας από το 2000 ίσα ίσα το βλέπει ως συμπληρωματική προσπάθεια ε, προς τις προσπάθειες του ΝΑΤΟ. Και εμείς όλα αυτά δεν τα κάνουμε για να ικανοποιήσουμε ε, τις επιθυμίες ε, των Αμερικανών φίλων που ζητούν από τους Ευρωπαίους να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες ή να αναλάβουν να σκόσουν το σταυρό τους. Δεν χρειάζεται να μας τα πούνε οι Αμερικανοί. ίδιοι οι πολίτες μας ζητούν να απαντήσουμε σε αυτές τις προκλήσεις που μπορεί να προέρχονται από ανατολικά ή από τον νότο. Βλέπουμε τι προσπάθειες έχει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα. Μία από τις μεγάλες μου ανησυχίε είναι η ζώνη ασφαλείας, όπως τη λέω, από την ε, Μαυριτανία μέχρι τη Σομαλία, για να μην μιλήσουμε για τη Λιβύη. Όλη αυτή λοιπόν η περιοχή και όλα τα θέματα είναι κάτι που δεν καλύπτει το ΝΑΤΟ, για να μην πω ότι δεν μπορεί να κάνει το ΝΑΤΟ για διάφορους λόγους τώρα. Δεν είναι ότι δεν ε, έχει τις τεχνικές δυνατότητες τις οποίες διαθέτει, αλλά για διάφορους λόγους η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να δράσει εκεί. Και είναι πιο πρόσφορη η δομή για να το κάνει. d'actions conjointes, mais au-delà des actions conjointes, on a Πέρα λοιπόν από τις κοινέ αυτές δράσεις, έχουμε αναπτύξει μια δυναμική συνεργασία και διαλόγου που στο παρελθόν δεν υπήρχε. Επαναλαμβάνω, αυτό το κάνουμε για να ικανοποιήσουμε κανέναν εξωτερικό, αλλά τις ίδιες μας ανάγκες και επιθυμίες και αιτήματα των πολιτών μας. Έτσι προσπαθούμε να ανταποκριθούμε σε αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much indeed. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρέσβη, για τις απαντήσεις που δώσατε στις ερωτήσεις μας. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται να εξαντλήσουμε ε, την ώρα που έχετε στη εσείς, γιατί έχετε και άλλη δουλειά. Ευχαριστώ που ήρθατε να μας ενημερώσετε και προσβλέπουμε και σε μελλοντική συνεργασία μαζί σας για να μας ενημερώνετε και να μας απαντάτε έτσι τόσο εκτενώς στις ερωτήσεις μας. Ευχαριστώ στο καλό. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, όπως ε, λοιπόν είχα ανακοινώσει στην αρχή της ε, συνεδρίασης, ε, πρέπει να κάνουμε ένα διάλειμμα για καφέ. Μέχρι τις 10 η ώρα ακριβώς, Δυστυχώς ε, δεν μπορούμε να επιταχύνουμε τις ε, διαδικασίες. Ε, έχουμε οργανώσει μια κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και βεβαίως θα συμμετέχουν και οι σχετικές αντιπροσωπείς. Το θέμα μας είναι η Βόρειος Κορέα. Παραμείνετε λοιπόν, γιατί θεωρούμε ότι θα έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες. Διάλειμμα μέχρι τις 10 ακριβώς παρακαλώ. Ευχαριστώ.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

Αγαπητοί συνάδελφοι, καλώς ήρθατε στην ε, ακρόαση μεταξύ, από κοινού οργανωμένη μεταξύ ε, Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Υποεπιτροπής Ασφάλειας ε, για την, το πυρηνικό πρόγραμμα της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας, γιατί υπήρξαν πολλές συζητήσεις για το θέμα αυτό κατά τους τελευταίους μήνες λόγω της σοβαρής απειλής για την ε, ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ειρήνη. Ε, είναι εδώ η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και προσκεκλημένοι οι οποίοι θα συμβάλλουν στην ε, συζήτησή μας για τη στρατηγική αυτής της κρίσιμης εμπλοκής στην από πυρηνικοποίηση της ε, ε, Βόρειας Κορέας ε, επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολλά να προσφέρει στην ανθρωπιστική βοήθεια που μπορεί να προσφέρει αλλά και στην οικονομική συνεργασία με την Βόρεια Κορέα. Ε, η ύπατη εκπρόσωπος και αντιπρόεδρος Φεντερίκα Μοντγκερίνη έπρεπε να αναλάβει ένα πολύ σημαντικό ρόλο ε, ως διαμεσολαβητής για να μπορέσουν να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ε, θα προετοιμάζει μια επίσκεψη στην Νότια Κορέα και στην Ιαπωνία στους στρατηγικούς εταίρους μας τον Απρίλιο του 2018 για να δείξει την υποστήριξη υπό το φως της νέας αυτής απειλής και ανταλλαγή απόψεων για το θέμα αυτό. Θα ήθελα να σας ε, δώσω το λόγο, να δώσω το λόγο στην ε, πρόεδρο ε, της Υποεπιτροπής Ασφάλειας, Άννα Φωτίγκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η αποστολή της Επιτροπής μας το Μάιο Ε, είχε ως στόχο την ε, συζήτηση ε, αυτήν την απειλή, την πυρηνική απειλή από τη Βόρεια Κορέα με τους εταίρους μας της περιοχής. Ήταν μια αποστολή στην Ιαπωνία και έγιναν συζητήσεις με πολλούς υψηλού επίπεδου συνομιλητές και για το θέμα αυτό. Βέβαια η ανώτατη, η ανώτερη στρατιωτική ηγεσία συμμετείχε επίσης ε, της Ιαπωνίας και ε, της Νότιας Κορέας και μετά από τις συζητήσεις αυτές μπορούσαμε και εμείς ε, να κάνουμε πολλές συζητήσεις. Ακούσαμε τις απόψεις των εταίρων της περιοχής Μετά τα εισαγωγικά μου αυτά σχόλια θα ήθελα να σας κάνω κάποιες τεχνικές παρατηρήσεις ε, πριν σας παρουσιάσω τους ομιλητές μας για την δημόσια αυτή ακρόαση. Όπως βλέπετε, είναι κοινή οργάνωση μεταξύ της Επιτροπής μας και της Υποτροπής Εξωτερικών ε, Υποθέσεων και έχουμε πολλούς προσκεκλημένους. Υπάρχουν και πολλές αντιπροσωπείες ε, των περιοχών των χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας ε, ε, με την, ε, της, της των σχέσεων με την Ιαπωνία, τη λαϊκή δημοκρατία της Κίνας και η αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Χερσόνησο της Κορέας. Συνάδελφοι, το τελευταίο, η τελευταία μας παρουσίαση θα γίνει μέσω Skype με τη Φλόριντα. Υπάρχει και διαφορά ώρας όπως γνωρίζετε. Δεν ε, θα είναι ένα δύσκολο πείραμα και για τους διερμηνείς. Δεν ξέρουμε για την ώρα αν έχουμε... Α, να, μπορούμε τώρα να δούμε τον κύριο Χίλ. Ε, καταφέραμε να έρθουμε σε επαφή μαζί του. Δεν τα είχαμε καταφέρει ως τώρα. Καλημέρα σας. Κυρίες και κύριοι, εξέχουσες προσωπικότητες σήμερα στο πάνελ μας. Να σας κάνω λοιπόν μια παρουσίαση των προσκεκλημένων μας που θα συζητήσουμε μαζί τους τις απειλές αυτές ε, ε, του, από το πυρηνικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας ε, Πρώτος προσκεκλημένος μας και ο μιλητής μας είναι ο κύριος Ράινχολ Μπρέντερ, ο οποίος είναι ε, τμήματάρχης για την Ιαπωνία, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και τον Ειρηνικό εντός της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Μετά το λόγο θα λάβει ο δόκτωρ Αντουάν Μπουντάζ, ο οποίος ε, είναι εδώ εκ μέρους ε, Ε, του Ιδρύματος για τη Στρατηγική Έρευνα, ερευνητής. και επίκουρος καθηγητής στο Σιόν Σπο στο Παρίσι. Είναι εδώ επίσης ο κύριος Ραμόν Πατσέκο Πάρντο από το Ίδρυμα ε, Κορέας, ε, λέκτορ στο King's College του Λονδίνου. Και επίσης μέσω Skype ε, θα συνδεθούμε με τον πρέσβη Κρίστοφερ Χίλ, ο οποίος είναι, έχει πολύ μεγάλη πείρα ένας πάρα πολύ πεπειραμένος διπλωμάτης, ε, Αμερικανός, τεράστια εμπειρία ε, για την περιοχή. Ειδικότερα δηλαδή για την Κορεατική Χερσόνησο. Έχει διατελέσει επίσης ε, και πρέσβη στην Πολωνία. Καλημέρα σας. Θα ήθελα, χωρίς να χρονοτριβήσω άλλο, να δώσω το λόγο στον κύριο Ράινχολτ Μπρέντερ, εκ μέρους της ΑΕΔ. E Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ε, αγαπητοί πρόεδροι των Επιτροπών Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Άμυνας, αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι τιμή για μένα, εκ μέρους Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, ε, να σας παρουσιάσω την κατάσταση που αφορά στην λαοκρατική δημοκρατία της Κορέας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνεί με την υπόλοιπη διεθνή κοινότητα ότι εμείς επιθυμούμε μια κορεατική ήπειρο η οποία ε, θα είναι ελεύθερη από πυρηνικά όπλα. Αυτό προ όφελο όλων των Κορεατών και του υπόλοιπου κόσμου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταδικάσει απερίφραστα ε, την ε, πυραυλική δοκιμή, την τελευταία τη ε, Κορέα, γιατί θεωρεί ότι αυτό αποτελεί κατάφορη παραβίαση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλεία των Ηνωμένων Εθνών και των σχετικών ψηφισμάτων. Οι πράξει αυτέ αποτελούν μια σοβαρή απειλή στη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Μετά λοιπόν από δυόμιση μήνε, χωρί σε πυρηνική ε, δοκιμή ή εκτόξευση πυράβλου η Βόρεια Κορέα στις 28 Νοεμβρίου, ώρα Βρυξελών, εκτόξευσε άλλο ένα πύραυλο και με βάση τις αρχικές εκτιμήσεις επρόκειτο για διεπιρωτικό βαλιστικό πύραυλο, ως εκ τούτου πύραυλο με πολύ μεγάλη εμβέλεια. Ε, ε, εκτοξεύτηκε από μια περιοχή βόρεια της ε, πρωτεύουσας της Πον Γιάνγκ και δίνει σε μια απόσταση περίπου 950 χιλιόμετρων. Στο ανώτατο ύψος της τροχιάς του έφτασε στα περίπου 4.500 χιλιόμετρα πριν προσγειωθεί στη θάλασσα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ιαπωνίας. Σε κανονική πορεία ο πύραυλος θα έχει διανύσει μια απόσταση 10.000 μέχρι 11.000 χιλιόμετρων. Με άλλα λόγια, τόσο οι Ηνωμένε Πολιτείε, η πυροτική έκταση των Ηνωμένων Πολιτειών, όσο και η Ευρώπη βρίσκονται πλέον μέσα στην εμβέλεια της, ε, των πυράβλων ε, που μπορεί να εκτοξεύσει η Βόρεια Κορέα, η οποία είπε και δήλωσε ότι είναι πλέον σε θέση να πλήξει όλη την υπηρετική Αμερική, της, ε, όπως επίσης ε, και ότι η χώρα πλέον έχει φτάσει σε μια ιστορική στιγμή που έχει ολοκληρώσει το πυρηνικό της πρόγραμμα. Αυτή τη στιγμή ε, βεβαίως δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορεί η Βόρεια Κορέα να σμικρύνει τα πυρηνικά όπλα έτσι ώστε αυτά να ε, τοποθετηθούν σε έναν πύραυλο. όλα αυτά η χώρα θεωρείται ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι σε θέση να διασφαλίσει το ότι ε, οι διπυρωτικοί βαλιστικοί πύραυλοι θα μπορούν να επανέλθουν σε επίπεδη επιχειρησιακή τροχιά άθικτη στην ατμόσφαιρα. Ως εκ τούτου ε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Βόρεια Κορέα τους τελευταίους δυόμισι μήνες ενώ δεν προέβη σε δημόσιες προκλήσεις παρόλα αυτά συνέχισε το πρόγραμμα πυρηνικού εξοπλισμού και δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι στο μέλλον ε, θα πάψει να κάνει κάτι τέτοιο. Εκείνο λοιπόν το οποίο συνέβη στις 28 Νοεμβρίου είναι απλά το τελευταίο βήμα που ανέπτυξε η Βόρεια Κορέα στο πρόγραμμά της ε, εκτόξευσης ε, πυράβλων με πυρηνικό εξοπλισμό. Υπήρξε μια δραματική επιτάχυνση τα τελευταία χρόνια. Θέλω να σας επενθυμίσω ότι τρεις ε, από τις έξι πυρηνικές δοκιμές της χώρας από το 2006, τρεις λοιπόν έλαβαν χώρα τα τελευταία δύο χρόνια. Και η τελευταία το Σεπτέμβρη και έφτασε μάλιστα στο, στους 100, στα 100 κιλοτόνους που είναι ένα υπερβολικά μεγάλος, ένας όγκος τεράστιος, 10 φορές περισσότερος από ό,τι ήταν το Σεπτέμβριο του 2016. Παράλληλα, το βαλιστικό ε, πρόγραμμα έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Ε, έχουμε 24 εκτοξεύσεις ε, πυράβλων το 2016 και 20 εκτοξεύσεις ε, το 2016, 20 μάλιστα από τις αρχές αυτού του έτους. Η εκτόξευση του τελευταίου, τον τελευταίο, του τελευταίου πυράβλου τον Νοέμβρη και πάλι προκάλεσε τη διεθνή καταδίκη. Η ότι εκπρόσωπος, η κυρία Μογκερίνη, μέσω του εκπροσώπου της, αποκάλεσε αυτή την εκτόξευση περαιτέρω σοβαρή πρόκληση και σοβαρή απειλή για τη διεθνή κοινότητα. Ε, κατόπιν ακολούθησαν εκκλήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Βόρειο Κορέα να συμμορφωθεί χωρίς καθυστέρηση, πλήρως και χωρίς προϋποθέσεις ε, στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει ε, στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε τη χώρα να απόσχει από άλλες προκλητικές ενέργειες που θα μπορούσαν να αυξήσουν επιπλέον την ένταση σε παγκόσμιο και ακόμα και περιφερειακό επίπεδο. Και να πω επίσης ότι ο πρόεδρος Τραμπ ανέφερε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε θα χειριστούν την κατάσταση στη Βόρεια Κορέα, ενώ ο Υπουργό Εξωτερικών τη χώρα, ο κ. Τίλερσον, ανέφερε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε καταδικάζουν απερίφραστα την εκτόξευση πυράβλου από τη Βόρεια Κορέα. Σε μια έκτακτη συνεδρία του Υπουργείου Ασφαλεία, οι Ηνωμένε Πολιτείε κάλεσαν πάλι όλε τι χώρε να υποβαθμίσουν ή να διακόψουν τι σχέσει του με τη Βόρεια Κορέα. Ε, το μήνυμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αδιαμφισβήτητο η Βόρεια Κορέα οφείλει να εγκαταλείψει πλήρω το πρόγραμμα βαλιστικών ε, ε, πυράβλων ε, και οφείλει αυτό να το πράξει με ένα πλήρη επαληθεύσιμο και μετάκλητο τρόπο. Οφείλει επίση η Βόρεια Κορέα να επανέλθει στην συνθήκη της μη διάδοσης πυρηνικών όπλων και σε αυτά που προβλέπει ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας. Όλες αυτές οι ενέργειες που έχουν αναπτυχθεί από τη Βόρεια Κορέα προβάλλουν το ότι είναι απαραίτητο να διεθνοποιηθεί η συνθήκη περί απαγόρευσης πυρηνικών όπλων. Το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών 2375 της 11 η Σεπτεμβρίου ήταν ένα σημαντικό βήμα για να επιταθεί η ένταση προς το καθεστώς της Βόρειας Κορέας. Και όπως ενδεχομένως θα θυμάστε, ε, το ψήφισμα αυτό έπρεπε βέβαια να εγκριθεί από την Κίνα και τη Ρωσία, πράγμα που έγινε και αυτό ήταν μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε πάρα αυτά αυτό το ψήφισμα και ακολούθησε το παράδειγμα που είχε προηγηθεί σχετικά με κυρώσεις που είχαν επιβληθεί στη Βόρεια Κορέα μέσω ψηφίσματος και πάλι των εθνών. Εξάλλου, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε άλλο, άλλη μια δέσμη αυτόνομων μέτρων, συμπληρωματικά μέτρα προς αυτά που αποφάσισαν τα Ηνωμένα Έθνη. Αυτά τα αυτόνομα μέτρα προβλέπουν επέκταση της απαγόρευσης σε όλες τις επενδύσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε όλους τους τομείς. Τώρα πλέον είναι αδιανόητο και δεν μπορούν να γίνουν επενδύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Κορέα. Επίσης προσθέθηκαν ονόματα και οντότητες σε αυτούς τους αυτόνομους καταλόγους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, προβλέπεται και απαγόρευση ταξιδίου για κάποιους ε, για κάποια άτομα και οντότητες ε, περιόρισε το ποσό των προσωπικών εμβασμάτων ε, προς την Βόρεια Κορέα από άτομα που εργάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό για να διασφαλιστεί ότι ε, στην Βόρεια Κορέα θα φτάνουν λιγότερα έσοδα για να μην είναι δυνατόν να στηριχτεί το πυρηνικό πρόβλημα στα αυτόνομα μέτρα προβλέπεται επίση απαγόρευση όλων των εξαγωγών πετρελαίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση προ την Βόρεια Κορέα. Ε, το θέμα των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα αντιμετωπιστεί και συμφωνήθηκε ότι οι άδειε εργασία για υπηκόου τη Βόρεια Κορέα που εργάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα ανανεωθούν εξαιρουμένων των προσφύγων και άλλων που απολάβουν διεθνού προστασίε. Άρα δηλαδή σιγά σιγά ε, θα εκλείψουν το συντομότερο βέβαια ετών οι ε, πίκο βόρειε Κορέας που εργάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επιπλέον το ε, Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών ενέκρινε έναν επικαιροποιημένο κατάλογο πολυτελών προϊόντων για το οποίο υπάρχει πλήρη απαγόρευση εισαγωγών και εξαγωγών. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι οι κυρώσει Ευρωπαϊκή Ένωση προ τη Βόρεια Κορέα είναι οι πιο αυστηρέ που υπάρχουν. Το εμπόριο ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Βόρεια Κορέα κατ' ουσίαν έχει σταματήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης σε επίπεδο κρατών μελών έχουμε ενισχύσει τις προσπάθειές μας για να διασφαλίσουμε ότι τρίτες χώρες θα συμμορφωθούν πλήρως με τις κυρώσεις που έχουν αποφασίσει τα Ενωμένα Έθνη. Γι' αυτό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνθηκε σε μια σειρά κρατών στην Αφρική και την Ασία ζητώντας να στηρίξουν αυτές τις αποφάσεις των Ενωμένων Εθνών. Εμείς λοιπόν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε κάνει αρκετά σημαντικά όχι μόνο για να εφαρμόζονται τα ψηφίσματα, αλλά και για να στηρίξουμε αυτόνομες κυρώσεις και επίση και για να καλέσουμε χώρες να στηρίξουν και αυτές πλήρως και ανεπιφύλακτα τις κυρώσεις των Ηνωμένων Εθνών. Το μήνυμά μας λοιπόν είναι απόλυτα σαφές. Να υπάρχει πλήρης εφαρμογή των ε, ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών αυτά τα ψηφίσματα που αφορούν την Βόρεια Κορέα και αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για να ασκηθεί πίεση στο καθεστώς να επανέλθει η Βόρεια Κορέα στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων. Ο στόχος, οι κυρώσεις μάλλον δεν αποτελούν αυτό σκοπό, είναι ένα εργαλείο για να ενθαρρύνεται ο πολιτικός διάλογος και να παραμένουν ανοιχτοί δίευλοι για το διάλογο. Το είπε εξάλλου και η Πρόεδρος. Τον Ιούλιο αυτού του έτου. <clears throat> οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαίωσαν μια πολιτική κριτικής απόσταση απόστασης θα λέγαμε από την Βόρεια Κορέα προβλέπονται μέτρα για να σκεφτούν πίεση βεβαίως ε, διατηρείται κάποιος διάλογος διατηρούνται διεύλοι διαλόγου Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τα πεπισμένοι ότι η αποπυρηνικοποίηση ε, πρέπει να επιτευχθεί μέσα από ειρηνικά μέσα και μέσα από το διάλογο. Αυτό εξάλλου υπογραμμίστηκε για άλλη μια φορά από του αρχηγού κρατών και κυβερνήσεων κατά τη συνάντησή τους στι 19 η και 20 η Οκτωβρίου. Το να είναι κανεί ειρηνικό δεν σημαίνει ότι είναι αδύναμος και το να είναι ισχυρό δεν σημαίνει ότι πρέπει απαραίτητα να ακολουθήσει το στρατιωτικό δρόμο, γιατί δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε τέτοιου είδου περιπτώσει. Ε, η κριτική αυτή απόσταση δεν είναι ο σκοπό, όπω σα είπα, είναι ένα τρόπο για να εφαρμοστούν πλήρω τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών για να εγκαταληφθεί το πρόγραμμα ε, το βαλιστικό, των βαλιστικών πυράβλων και αυτό να γίνει όπω σα είπα με ολοκληρωμένο, επαληθεύσιμο και αμετάκλητο τρόπο. Εμεί παραμένουμε πρόθυμοι να συνεργαστούμε με όλου του άμεσα ενδιαφερόμενου για να ασχίσουμε τη μέγιστη οικονομική και διπλωματική πίεση που μπορούμε έναντι της Βόρειας Κορέας. Προσβλέπουμε ε, σε αυτά που θα ε, αναφέρει ο Τζέφρι Φέλτμαν, αναπληρωτής ε, γενικός γραμματέας από την επίσκεψή του στη Βόρεια Κορέα. Θέλουμε να δούμε κατά πόσον υπάρχουν στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν να ανοίξει μια διπλωματική λύση. Εξάλλου, εμείς θεωρούμε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιαπωνίας, ο κύριος Κόνο, θα ε, προεδρεύσει σε μια υπουργική συνάντηση στο Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ στις 15 Δεκεμβρίου για να συζητηθεί το πυρηνικό και βαλιστικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας. Την προηγούμενη εβδομάδα επιβεβαιώθηκε ότι οι ΗΠΑ και ο Καναδάς στις αρχές του επόμενου έτους θα ε, συμπροεδρεύσουν σε μια υπουργική συνάντηση για να συζητήσουν το πώς η διεθνής κοινότητα μπορεί να αντιμετωπίσει τις ε, προκλήσεις της Βόρειας Κορέας. Η ενότητα της διεθνούς κοινότητας στην αντιμετώπιση προκλήσεων του πυρηνικού και βαλιστικού προγράμματος της Βόρειας Κορέας είναι ένα στοιχείο καθοριστικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναζητήσει επαφέ με όλου του σημαντικού εταίρους τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή και αυτό το έχει πράξει μέσα από συγκεκριμένε ενέργειε, αλλά και μέσα από την ανεπιφύλακτη υποστήριξη όλων των κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών. Συνεχίζουμε τι σχέσει με του ε, εταίρους μα εντό και εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε συζητήσεις για το ποια είναι η η καλύτερη δυνατή αντίδραση στην τελευταία εκτόξευση βαλιστικών πυράβλων. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Ε, κύριε, θα δώσω τώρα το λόγο στον δόκτωρο Αντουάν ε, Μποντάζ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ε, αξιότιμη πρόεδρε, αντιπρόεδρε της Επιτροπής Εξωτερικών, αξιότιμη πρόεδρε της Επιτροπής ΕΔΕ, κυρίες και κύριοι ευρωβουλευτές, είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή ε, που αισθάνομαι να σας απευθύνω το λόγο. Στις 29 Νοεμβρίου η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας ανακοίνωσε ότι επιτέλους είχε την ιστορική ε, πραγματικότητα του να είναι πυρηνική δύναμη. Ε, την προηγούμενη ημέρα ε, ε, είχαν εκτοξεύσει ένα διεπηρετικό βαλιστικό πύραυλο Χουάσονγκ 15 που θα μπορούσε για πρώτη φορά να φτάσει σε οποιαδήποτε πόλη ε, στην επιρωτική Αμερική στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό πραγματικά εντάσσεται στη στρατηγική επιβίωση που έχει στόχο να ενισχύσει την αποτροπή αλλά και την εσωτερική νομιμοποίηση του Κιμ Ιονγκ Ουν και επίσης σηματοδοτεί μια νέα δυνατότητα διαπραγματεύσεων αν θέλουμε να κάνουμε ένα πρώτο βήμα προς την αποπυρηνικοποίηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ρόλο και ενδιαφέρον να παίξει αυτό το ρόλο. Τα δύο προγράμματα ε, δεν μπορούν να αποσυνδεθούν μεταξύ τους. Η Βόρεια Κορέα έχει ε, σκληρύνει τις τάσεις για τα πυρηνικά με τον νέο ηγέτη ήδη από το 2013 το έχει θέσει τεχνική προτεραιότητα, τη ε, την ελάφρυνση των πυράβλων, τη διαφοροποίησή τους και την αύξηση της ακρίβειάς τους. Επίσης, παρήγγειλε τέσσερις νέες πυρηνικές δοκιμές από το 2013 μέχρι το 2017 και μέχρι και θερμοπυρηνική ε, βόμβα. Δεύτερον, το καθεστώς άρχισε να θεσμοποιεί αυτά τα όπλα. Ε, η Ανώτατη Λαϊκή Συνέλευση, η πρόεδρος Ιακώπτη τον μήπως να μιλάτε λίγο πιο αργά, να διαβάζετε λίγο πιο αργά, γιατί οι διερμηνείς δεν σας προλαβαίνουν. Δεύτερον, ε, το καθεστώς έχει πλέον θεσμοθετήσει αυτά τα όπλα. Η Ανώτατη Λαϊκή Συνέλευση αναθεώρησε το Σύνταγμα στις αρχές του 2012 ε, ε, έτσι ώστε η χώρα να αναφέρεται ως πυρηνική δύναμη, πυρηνικό κράτος, το πρώτο στον κόσμο. Αυτή η εξέλιξη και η ανάπτυξη των πυρηνικών έχει εγγραφεί και στην Εθνική Στρατηγική που παρουσιάστηκε στις 31 Μαρτίου το 2013, η λεγόμενη Μπιουντζίν, που έχει στόχο ε, την οικονομική οικοδόμηση, την ανάπτυξη και δημιουργία ε, πυρηνικών ενόπλων δυνάμεων ταυτόχρονα. Ε, ήταν η εξέλιξη της πολιτικής του προηγούμενου ηγέτη με στόχο πρώτα τη στρατιωτική ισχύ. Από το 2013 αυτό έχει ενισχυθεί. Ο Κιμ Τζονγκούν έχει διατάξει 20 πυρηνικές δοκιμές μόνο το 2017 περισσότερες από τις 16 ε, δοκιμές που είχε διατάξει ο πατέρας του σε 15 χρόνια και συνολικά πάνω από 80 δοκιμές αφού του ανέλαβε καθήκοντα ο Κιμ Γιονγκούν. Στη συνέχεια ε, το καθεστώς έχει διαφοροποιήσει τους πυράβλους για πρώτη φορά ε, κάνει δοκιμές ε, για πυράβλους μεσαίου βεληνικούς Χουάσον 12 και διπυρωτικούς πυράβλους Χουάσον 14 και 15 το 2017. Είναι πύραυλοι που ε, δεν απειλούν μόνο συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ασία και τον Ειρηνικό, αλλά για πρώτη φορά και την επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Και τέλος, τοποθεσίες εκτόξευσης έχουν ε, πολλαπλασιαστεί, είναι πάνω από 15, ενώ επί Kim Jong-il ήταν μόνο δύο. Ε, τώρα επίσης εκπαιδεύονται και οι στρατιωτικοί για να έχουν και νυχτερινές δοκιμές δεν, δεν ε, δοκιμάζουν δηλαδή μόνο τα τεχνικά χαρακτηριστικά, αλλά προχωρούν και σε στρατιωτικές ε, δοκιμές. Ποιος είναι ο στόχος, σαφής, το συντομότερο να γίνει η πυρηνική δύναμη, η Βόρεια Κορέα, να είναι η αποτροπή της η πυρηνική πίστευτη, να ενισχυθεί η νομιμοποίηση του Κιμ Γιονγκούν και να ενισχυθεί ο, πι, ο ε, με τις Ηνωμένες Πολιτείες στις διαπραγματεύσεις. Αυτό εντάσσεται στη στρατηγική επιβίωση του καθεστώτος προς τα έξω αλλά και προς το εσωτερικό της χώρας. Η εξωτερική διάσταση έχει σχέση με την ασφάλεια του καθεστώτος από εξωτερικές απειλές. Τα πυρηνικά όπλα ε, καταπραίνουν λίγο την παράνοια της Βόρειας Κορέας και τους καθεστώτος σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την εχθρική πολιτική τους και τις πυρηνικές απειλές. Όλα αυτά είναι παραθέσεις. Ε, το γεγονός ότι η Βόρεια Κορέα θα έχει πυρηνικά όπλα ε, αυξάνει το επίπεδο αποτροπής που είναι αρκετά υψηλό ε, γιατί επί δεκαετίε ήταν όμοιρο των συμβατικών δυνατοτήτων. Η εσωτερική διάσταση είναι ακόμα πιο σημαντική και έχει να κάνει με την σταθερότητα του καθεστώτος από εσωτερικές απειλέ. Τα πυρηνικά όπλα είναι πολιτικά όπλα που ενισχύουν την ομιμοποίηση του Κιμ Τζονγκούν και την παραμονή του στην εξουσία. Πρώτα, ε, εδρεώνουν το ε, σύστημα, το κληρονομικό της εξουσίας. Ε, δεύτερον, αυξάνουν το κύρος του ως προστάτη του ε, κορανικού ε, κορεατικού συγγνώμη, έθνους που έχει φέρει ασφάλεια στο λαό του, ένα μεγάλο επίτευγμα που συνεχίζει την παράδοση του παππού του και του πατέρα του. Τρίτον, νομιμοποιούν τις δεκαετίες θυσιών για να στηθεί αυτό το καθεστώς τέταρτο και τελευταίο ενισχύουν την εσωτερική συνοχή και ε, το ηθικό του έθνους. Όπως φαίνεται ε, και φάνηκε την 1η Δεκεμβρίου από τις μαζικές διαδηλώσεις. Επίσης, ε, τα πυρηνικά ταυτίζονται με το Τζούντζε, την ιδεολογία που έχουν, ε, την εθνολαϊκή. Ε, αναζητούν πολιτική ανεξαρτησία για αυτόνομη οικονομία και δυνατότητα αυτοάμυνας. Ε, η κατοχή πυρηνικών όπλων είναι πρωτοφανής πηγή νομιμοποίησης γενικά για ένα καθεστώς που σύμφωνα με την προπαγάνδα του είναι υπέρ της ανεξαρτησίας και της αυτονομίας της Κορέας μετά από αιώνες ε, ξένης επιρροής και ξένης κατοχής. Τώρα είναι απαραίτητο εργαλείο για την πολιτική εφαρμογή του Τζούντσε, του συστήματος του καθεστώτος και η θεσμοθέτηση των πυρηνικών ε, είναι ένα τμήμα της ε, ταυτότητας του καθεστώτος. Δεν είναι απλώς ότι έχει κατοχή πυρηνικών όπλων. και δεν αμφισβητείται από το εσωτερικό ε, πλέον ο Κιμ Ιονγκ Ουν. Και είναι σε θέση ένας νέος ε, ηγέτης να ανακοινώσει ότι έχει ολοκληρώσει την πυρηνική προσπάθεια και μπορεί να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις. Το θέμα ε, είναι τώρα η διεθνή κοινότητα να αποτρέψει την ανάπτυξη πυρηνικών και βαλιστικών πυράβλων. Είμαστε σε ένα σταυροδρόμι και είναι προτεραιότητα να παραμείνει η αξιοπιστία του ΟΗΕ και της διεθνούς κοινότητας με την εφαρμογή και το σεβασμό από όλου των αντιστοίχων ψηφισμάτων. Δεν ακούν οι κυρώσεις από μόνες τους. Υπάρχει ένα πάνελ του ΟΗΕ 17-18 που δείχνει ε, ότι η Κορέα περιφρονεί τις ε, κυρώσεις και με διάφορους τρόπους τις παρακάμπτει. Επίσης, δεν υπάρχει και αντίστοιχη πολιτική βούληση. Ούτε χρησιμοποιούν τους σπόρους που χρειάζεται για να τα εφαρμόσουν ε, πλήρως. Έχουμε ψηφίσματα 2371 μέχρι 2375 που αναφέρονται ε, για στις κυρώσεις, αλλά δεν πρόκειται να αλλάξει ε, τη στάση του καθεστώτος, γιατί θεωρεί το καθεστώς ότι υπάρχουν πολιτικά και στρατιωτικά ωφέλη από το πυρηνικό πρόγραμμα πολύ μεγαλύτερα από το οικονομικό και το διπλωματικό κόστος που ενέχουν. Αλλά είναι πάρα πολύ νωρί να πούμε ότι έχουν αποτύχει οι κυρώσεις, γιατί οι οικονομικές κυρώσεις έχουν αρχίσει μόλις φέτος. Η χρησιμότητα των κυρώσεων θα αξιολογηθεί μετά την πλήρη εφαρμογή τους ε, ε, ως ευρύτερη στρατηγική. Ε, υπάρχουν στρατιωτικές κυρώσεις, ε, μπορεί να αποτρέψουν τη Βόρεια Κορέα, αλλά δεν θα την ε, αναγκάσουν σε κανένα βαθμό να αποστεί του πυρηνικού προγράμματος. Υπάρχει κόστος πολιτικό, ε, οικονομικό και ανθρώπινο, αφόρητο και οι πιθανότητες επιτυχίας είναι πολύ μικρές. Αφήστε δε που οι στρατιωτικές επεμβάσεις και οι βομβαρδισμοί δεν πρόκειται να αποδυναμώσουν το καθεστώ ούτε να καταστρέψουν εγκαταστάσει, γιατί οι περισσότερε είναι υπόγειες. Ε, και θα χρειαστεί ε, οπωσδήποτε ε, επέμβαση ειδικών δυνάμεων ε, χερσαίων. Ένας πόλεμος, ακόμα και συμβατικός, θα είχε τεράστιες επιπτώσεις. Υπάρχουν χιλιάδες Ευρωπαίοι και 300.000 Αμερικανοί και 60.000 Ιάπωνες που ζουν στη Νότια Κορέα. Επίσης, θα μπορούσε να, με κάποιο τρόπο να εμπλακεί η Κίνα για να τους βοηθήσει, γιατί έχουν σύμφωνο αμυντικό από το 1961. Και ο οικονομικός αντίκτυπος στα χρηματιστήρια και στο εμπόριο θα ήταν τεράστιος. Γιατί ένας τέτοιος πόλεμος ε, θα ξεσπούσε στον ίδιο τον κινητήρα της παγκόσμιας οικονομίας. Η σταθερότητα λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνδέεται με τη σταθερότητα στην Κορεατική Χερσόνησο, γιατί αν ε, χρησιμοποιηθεί η ε, πολεμική απειλή, τότε αυξάνεται ο κίνδυνος ε, σφάλματος, λάθος εκτίμησης, ενώ ο στόχος της διεθνούς κοινότητας είναι η αποπυρηνικοποίηση. Ένας στόχος καθαρός και βραχυπρόθεσμος θα μπορούσε να είναι συγκράτηση της απειλής, πριν βελτιώσει ακόμα περισσότερο τις δυνατότητές του το καθεστώς. Δηλαδή ένα πάγωμα του προγράμματος με ενίσχυση δράσεων για την πρόληψη της διάδοσης και την ε, αποφυγή των κυρώσεων. Αυτό το πάγωμα πρώτα θα σταματήσει την ανάπτυξη της τεχνολογίας και μετά θα την ε, καταστρέψει. Το 2010 υπήρξε μια συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Βόρειας Κορέας, άρα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ε, αναγνώρισή τους ως πυρηνική δύναμη. Ταυτόχρονα περιορίζεται η απειλή, ενώ στη συνέχεια θα υπάρξουν διαπραγματεύσεις για την περαιτέρω αποπυρηνικοποίηση. Επιπλέον και οι Ηνωμένε Πολιτείε αλλά και η Βόρεια Κορέα μπορούν να έρθουν στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων από θέση ισχύω. Η Βόρεια Κορέα λόγω της τεχνικής προόδου, ενώ οι Ηνωμένε Πολιτείε χαιρούν τη υποστήριξη τη διεθνού κοινότητα. Η υποστήριξη τη Κίνα είναι επίση σημαντική, αλλά θα πρέπει να συζητήσουμε και ε, ε, την ε, Συνορωσική Συμφωνία για το πάγωμα των λεγόμενων αγαθών διπλής χρήσεως. Ε, για κάποιες καταστάσεις που είναι απαράδεκτες για τις ΗΠΑ και τους συμμάχους. Τελευταία σημεία. Χρειάζεται ε, καλύτερη εφαρμογή των κυρώσεων και καταπολέμηση των ε, παρανόμων δραστηριότητων της Βόρειας Κορέας στην Ευρώπη και καλύτερη βοήθεια των εταίρων μας στην Ασία, την Αφρική και την Μέση Ανατολή, όπως είπε ο κύριος Μπρέντερ. Δεύτερον, πρέπει να σφυριλατηθεί ένας διάλογος με τη Βόρεια Κορέα και να διευκολυνθεί ο διάλογος μεταξύ των ε, πρωταγωνιστών και μεταξύ Βόρειας Κορέας και Ηνωμένων Πολιτειών κυρώσεις και διάλογος πρέπει να συμβαδίζουν. μέγιστη πίεση και διάλογος. Αυτά αποδίδουν. Διάλογος μεταξύ των μερών. Αυτό παραμένει ζωτικό για να καταλάβουμε ε, τις προθέσεις τους και να πείσουμε το καθεστώς ότι σε περίπτωση που αλλάξει τακτική και σεβαστεί ε, το ε, διεθνές δίκαιο θα έχει ωφέλη. θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και την πρόσβαση που έχει η Ευρώπη εκεί, ενώ η Αμερική, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα ε, δεν έχουν. 64 χρόνια μετά τον πόλεμο της Κορέας, τεχνικά η Κορεατική Χερσόνησος είναι σε εμπόλεμη mm. φάση. Θα μπορούσαμε να προτείνουμε την υπογραφή νευτικής συμφωνίας ε, ταυτόχρονα με την αποπενικοποίηση της Βόρειας Κορέας. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Now, Dr. Ramon Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δίνω το λόγο τώρα στον Ραμόν Πατσεκοπάρδο από το King's College του Λονδίνου. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση προκειμένου να συμμετάσχω στη σημερινή ακρόαση. Ε, πρόεδροι των Επιτροπών ε, ε, Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής, Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας. Έχω προετοιμάσει κάποιες διαφάνειες που θα τις χρησιμοποιήσω ως γνώμονα για την παρουσίασή μου. <laughs> Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Μου ζητήθηκε να ε, επικεντρωθώ στις ε, στρατηγικές πτυχές, στις ε, απειλές και στις πιθανές λύσεις για τις, στην πυρηνική αυτή κρίση της Βόρειας Κορέας. Θα επικεντρωθώ λοιπόν στις απειλές, αλλά πιο σύντομα, γιατί οι προηγούμενοι ομιλητές ε, το κάλυψαν αυτό το θέμα, νομίζω πολύ καλά. Ε, μετά θα εστιάσω στις στρατηγικές ε, διαστάσεις, όπως επίσης και στο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά τη γνώμη μου, έχει καταστεί πιο σημαντικός παίκτη στην ενδεχόμενη λύση της επίλυση της πυρηνικής αυτής κρίσης, της προερχόμενης από τη Βόρεια Κορέα. Οι προηγούμενοι ομιλητές μίλησαν για αυτή την άμεση πυρηνική απειλή του πυρηνικού προγράμματος της Βόρειας Κορέας για την Νότια Κορέα, οπότε δεν θα αναφερθώ σε αυτό. Επίσης αναφέρθηκε πολύ το γεγονός ότι φαίνεται ότι, δεν είναι, ότι, ότι υπάρχει η, πιθανότητα ε, ε, ε, να υπάρξουν πλήγματα για τις Ηνωμένε Πολιτείες, την Ιαπωνία και την Νότια Κορέα. Δεν θα το αναφέρω αυτό διεξοδικότερα. Ε, υπάρχει όμως ένα σύνολο περιφερειακών προγραμμάτων, προβλημάτων που έχουμε στην Νότιο Ανατολική Ασία. Όπως γνωρίζετε για παράδειγμα στην Ανατολική Θάλασσα ή Θάλασσα η Ιαπωνική, Ιαπωνική Θάλασσα, ε, ε, αναφέρομαι ε, στα διαφιλονικούμενα νησιά που υπάρχουν εκεί. Ε, υπάρχει περίπτωση ε, να χρησιμοποιηθεί η στρατιωρική απειλή ε, αν ε, η Ιαπωνία θέλει να πάρει πίσω αυτά τα νησιά που τώρα αυτή τη στιγμή ανήκουν στην Νότια Κορέα. Υπάρχει αυτή η ιδέα του τι θα συμβεί αν υπάρξουν, αν, αν συζητηθούν μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών αυτό το μεγάλο η συμφωνία για την Ταϊβάν ε, είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει επίσης να το ξεχνάμε. Ναι. Κύριε Πατσεκοπάρντο, θέλω να σας ζητήσω, λέει η πρόεδρο, να μιλάτε λίγο πιο αργά. Ναι, ξέρετε, οι Ισπανοί μιλάμε πολύ γρήγορα. Θα ήθελα να εστιαστώ ε, στο καθεστώς μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, ε, κάτι το οποίο δεν συζητήθηκε. Όπω γνωρίζετε, η Νότια Κορέα ε, στο παρελθόν έχει κάνει μια διάδοση όπλων στη Λιβύη, στην Αίγυπτο, στο Ιράν. Έχουν επωφεληθεί αυτέ οι χώρε από μετάδοση ε, γνώσης ε, και υλικού. Είναι μια απειλή λοιπόν όχι μόνο στην Νοτιοανατολική Ασία αλλά και σε αυτήν την περιοχή, η οποία είναι πολύ κοντά γεωγραφικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό τι θα γίνει για παράδειγμα αν άλλες πυρηνικές ε, δυνάμεις ε, ενθαρρυνθούν από το ότι μπόρεσε η Βόρεια Κορέα να αναπτύξει το πυρηνικό της πρόγραμμα. Ε, υπάρχει ας πούμε τώρα μια αμφιβολία για την ε, συμφωνία με, την, με το Ιράν, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και το Ιράν. Τι θα γίνει αν οι Ηνωμένε Πολιτείε αποσυρθούν από αυτήν τη συμφωνία και ακολουθήσει το Ιράν την ίδια πορεία με τη Βόρεια Κορέα. Να σας επιστήσω επίσης την προσοχή ότι έχουμε πάρα πολύ συζητήσεις και στην Νότια Κορέα και στην Ιαπωνία σε σχέση με την ανάπτυξη των δικών τους πυρηνικών προγραμμάτων. Για την ώρα στην Νότια Κορέα έχουν εστιαστεί στην εκ νέου ανάπτυξη τακτικών όπλων ε, από τις ΗΠΑ, αλλά, ε, μέχρι, αλλά περίπου δύο τρίτα των ε, ε, ε, πολιτών της Νότιας Κορέας υποστηρίζουν το πυρηνικό πρόγραμμα. Αν λοιπόν η Ιαπωνία κάνει το ίδιο, που μπορεί να είναι μικρότερη υποστήριξη, 23%, ε, υπάρχει δυνατότητα μιας, ενός πυρηνικού καταμερισμού με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Δηλαδή η Ιαπωνία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τις πυρηνικές ικανότητες των Ηνωμένων Πολιτειών αν, θεωρηθεί ότι, αν θεωρήσει ότι απειλείται από τη Βόρεια Κορέα. Δεν λέω ότι θα γίνει αυτό σύντομα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πολύ ανοιχτέ οι συζητήσεις ε, και μπορούν να, ε, μπορείτε να τις παρακολουθείτε και εσείς εδώ ε, στην Ευρώπη. Πρέπει να επικεντρωθούμε επίσης και στις περιφερειακές στρατηγικές ε, ε, διαστάσεις αλλά και στις παγκόσμιες στρατηγικές διαστάσεις του προβλήματος. Αυτός ο ανταγωνισμός μεταξύ της Βόρειας και της Νότιας Κορέας, μην ξεχνούμε ότι υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ τους για την νομιμοποίηση. Είναι προφανές ότι για οικονομικούς, διπλωματικούς λόγους είναι πιο νομιμοποιημένη χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο η Νότια Κορέα αλλά η Βόρεια Κορέα θεωρεί ότι το πυρηνικό της πρόγραμμα είναι ένα πλεονέκτημα συγκλητικό σε σχέση με την ε, Νότια Κορέα, γιατί η Νότια Κορέα δεν έχει πυρηνικά όπλα. Τι κάνει λοιπόν αυτή τη στιγμή η Νότια Κορέα, αυξάνει τη στρατιωτική της ικανότητα του χρόνου, για παράδειγμα, ε, θα έχει ένα, ένα, μία, θα έχει ένα πρόγραμμα μη επανδρομένων ε, ε, αεροσκαφών, drones. θα το αυξήσει, θα το ενισχύσει αυτό το πρόγραμμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης δεν δίνουν πια όρια ως οι Ηνωμένε Πολιτείες δεν Ε, ε, είναι λοιπόν πάρα πολύ δύσκολο γιατί οι Ηνωμένε Πολιτείε και αυτέ έχουν αρχίσει τα όρια να ε, τα, μετακινούν κάπω. αν οι όταν, κάποιο, όταν επειδή υπήρχε, υπήρχαν διπλωματικές σχέσεις μεταξύ της Κίνας και της Βόρειας Κορέας, μετά το πυρηνικό πρόγραμμα ε, αναφέρθηκε ότι ε, αυτό είναι το τέλος των διπλωματικών σχέσεων. Ε, το θέμα είναι κατά πόσο μπορούμε να προσπαθήσουμε να υπάρχουν κάποιες διαπραγματεύσεις. είναι κάτι το οποίο το έφεραν και οι συνάδελφοι προηγουμένως. Πλέον Υπάρχουν περισσότερες κυρώσεις ε, για την Βόρεια Κορέα μετά την πυρηνική αυτή ε, εξέλιξη το θέμα είναι πόσο οι Ηνωμένε Πολιτείε παραμένουν αφοσιωμένες στις συμμαχίε τους. Αν υπάρξει ε, επίθεση από τη Βόρεια Κορέα θα είναι σε θέση να αντεπιτεθούν ή να υποστηρίξουν την Νότιο Κορέα. Για παράδειγμα, η απάντηση μπορεί να υποστηριξουν τη νοτιο κορεα για παραδειγμα η απαντηση μπορει να ειναι ναι, αλλά όταν βλέπετε τη συζήτηση στο πλαίσιο της ε, Ιαπωνίας και της νότια Κορέα για, για τη δέσμευση αυτή, το, το ζήτημα της στρατιωτικοποίησης γίνεται πολύ πιο σοβαρό και στις δύο χώρες. υπάρχει λοιπόν αυτή η συζήτηση για το άρθρο 9 του συντάγματος και τη στρατιωτικοποίηση. Ε, η Ιαπωνία για παράδειγμα τώρα συζητά ανοιχτά και ίσως την επόμενη χρονιά να το κάνει, να αποκτήσει πυράβλους ε, που μπορούν να επιτεθούν στη Βόρεια Κορέα. Η Ιαπωνία για την ώρα δεν έχει αυτή την ικανότητα θεωρητικά, αλλά του χρόνου μπορεί να την έχει. Οπότε αυτό το θέμα της στρατιωτικοποίησης και όχι μόνο της πυρηνικοποίησης είναι ε, παρόν. Σε παγκόσμιο επίπεδο τώρα έχουμε αυτό το σημείο ανάφλεξης από απόψεω ασφάλεια. πρέπει να συζητούμε την Βόρεια Κορέα συνεχώς στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Πρέπει να το συζητούμε ε, στην Νοτιοανατολική Ασία. Υπάρχουν ε, οικονομικές συνέπειες που αναφέρθηκαν εν μέρη προηγουμένως. Ε, υπάρχει λοιπόν αυτό το ζήτημα το συνεχές ασφαλείας στην περιοχή. Το είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητέ. Μέχρι τώρα οι κυρώσει δεν έχουν υπάρξει αποτελεσματικές. Ε, ε, ε, άρχισαν το 2006. 11 χρόνια μετά η Βόρειος Κορέα έχει ένα πλήρες πυρηνικό πρόγραμμα και μπορεί να υπάρχουν και άλλες χώρες οι οποίες μπορεί έτσι να θεωρήσουν ότι και εκείνες καλά θα κάνουν να αναπτύξουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα όχι de jure, αλλά εν πάση περιπτώσει μια de facto αναγνώριση της πυρηνικής ε, δύναμης ε, της Βόρειας ε, Κορέας. Μερικές φορές θεωρείται ε, μάλλον συζητιέται τι θα είχε γίνει αν το Ινδία και το, το Πακιστάν είχαν ε, όντω και εκείνε αναγνωριστεί όπω είχε γίνει και γιατί να μην συμβαίνει για το ίδιο και με τη Βόρεια Κορέα. Όμω οι λόγοι είναι διαφορετικοί και η, το πλαίσιο είναι διαφορετικό. Η, ίδια η Βόρειο Κορέα λέει στο Σύνταγμά τη ότι είναι πυρηνικό κράτο πλέον. Θα ήθελα να επικεντρωθώ επίση στι ε, πιθανέ λύσει για το μετριασμό και την ανάσχεση. Είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ περίπλοκο. Διαφορετικά θα το είχαμε λύσει ήδη. Αν επικεντρωθούμε στη Βόρεια Κορέα, νομίζω ότι είναι βασικό ο διάλογο και μιλάω για τον επίσημο διάλογο. Υπάρχει ανεπίσημο διάλογο που γίνεται μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και ε, Βόρεια Κορέα. Όμω ο επίσημο διάλογο είναι και αυτό απαραίτητο. Θέλει αναγνώριση, είναι τμήμα τη αναγνώριση ω ε, κανονικό παίκτη ε, ε, στο διεθνέ προσκήνιο. Χρειαζόμαστε μία επίσημη δέσμευση ε, επίσης αυτό έρχεται σε αντίθεση με αυτό που λέει συνήθως ότι είναι απομονωμένη η Βόρεια Κορέα, επομένως πρέπει να αναπτύξει τις δικές της αμυντικές ικανότητες. Νομίζω ότι η εμπλοκή και άλλα είδη εμπλοκής, εκτός της οικονομικής, είναι απαραίτητα. γιατί όπως είπαμε προηγουμένως ε, η οικονομία και η στρατοικοποίηση για αυτή τη χώρα πηγαίνουν μαζί και αν πάμε πίσω στον Ιούλιο του 2002, βλέπουμε ότι από τότε έχει μπει σε μια διαδικασία οικονομική μεταρρύθμιση που ακολουθεί κατά κάποιο τρόπο το μοντέλο του Βιετνάμ και τη Κίνα, αλλά είναι πιο κοντά στο Βιετνάμ, θα έλεγα, ε, λόγω του μεγέθου τη χώρα. Δεν μπορεί να συγκριθεί με την Κίνα από απόψεω μεγέθου. Θα ήταν χρήσιμο λοιπόν αν η Βόρεια Κορέα προσπαθεί να αναπτύξει ε, κάποιους οικονομικούς τομείς, ε, την ενδυμασία, τη στέγη. Χρειάζεται να γίνει κάτι τέτοιο. Όσον αφορά τώρα τη μη διάδοση, πώς είναι δυνατόν να μετριάσουμε και να ε, κάνουμε ανάκριση αυτής της απειλής... Ε, Κάποιε κυρώσει χρειάζονται, δεν μπόρεσαν να παρεμποδίσουν βέβαια την ανάπτυξη του προγράμματο. Ε, Παρ' όλα αυτά είναι ένα ισχυρό μήνυμα. Να πάω πίσω ε, στο 2005 και στι ε, συζητήσει που έγιναν μετά τη συμφωνία τότε. Ε, τις εξαμερείς συμφωνίες θέλουμε να, κάνουμε μια σταδια... να υπάρχει μια σταδιακή προσέγγιση μείωση τη απειλή. Κάποιες κυρώσεις θα μπορούσαν να μειωθούν ώστε να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Όσον αφορά όμως μη διάδοση κάτι που συχνά ξεχνούμε αλλά ήταν επιτυχές, ήταν ε, η πρωτοβουλία ασφάλειας κατά της διάδοσης ε, όσον αφορά την πυρηνική τεχνολογία και τα, μέσα, τα όπλα μαζικής καταστροφής που έχουν μειωθεί. Όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετέχουν σε αυτήν την ε, πρωτοβουλία. Η υπάρχουν ε, τελωνιακοί έλεγχοι που γίνονται, υπάρχουν κυρώσεις ε, για τις εταιρείες που λειτουργούν ε, και συναλλάσσονται και με τη Βόρεια Κορέα. Νομίζω ότι τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες είναι απαραίτητες και πρέπει να συνεχίσουν. Και πάμε στο τελευταίο κομμάτι της παρουσίασής μου, το οποίο αφορά το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα μπω σε πάρα πολλέ λεπτομέρειε. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει. Πρώτον, να υποστηρίξει και να συντονίσει την, ε, το διάλογο και μαζί με άλλους ε, εταίρους. Η διπλωματική υποστήριξη συχνά είναι πολύ σημαντική και μπορώ να σας πω ότι στη Νότια Κορέα είχε σημαντικό ρόλο όταν είχε πει ε, στο καθεστώς ότι θα έπρεπε να συμμετέχει πιο ενεργά στην επίλυση του πυρηνικού προβλήματος λόγω της, του πυρηνικού προγράμματος της Βόρειας Κορέας. Επίσης, ε, η διαμεσολάβηση στην Νοτιοανατολική Ασία Βόρειο Ανατολική Ασία, συγγνώμη, ε, είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι θεσμοθετημένη μάλιστα. Ε, η Ρουμανία, η Πολωνία, η Σουηδία, η Γερμανία έχουν πληροφορίες επιτόπου σε σχέση με το τι συμβαίνει που άλλε χώρε δεν έχουν στη διάθεσή του, οπότε η συνεργασία είναι πολύ σημαντική και θα έπρεπε να υπάρχει και υποστήριξη για την επίσημη οικονομική υποστήριξη, ε, εκπαίδευση από την Νότια Κορέα και από άλλες χώρες, ε, συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, ε, πολιτικές, αθλητικέ ανταλλαγές και μερικές φορέ. και επιχειρηματικές αναλλαγέ, γιατί μπορεί να διαμορφώσουν τη συμπεριφορά της ε, Βόρειας Κορέας και αν υπάρχει πολυμερής διάλογος τελικά, νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πιέσει ε, το, ε, να, συμμετοχή στο διάλογο ή να την υποστηρίξει το Ηνωμένε Πολιτείε μπορεί να μην συμμετέχουν, αλλά ε, στο παρελθόν η Ευρωπαϊκή Ένωση το είχε κάνει, συμμετείχε ε, στην, ε, στο πλαίσιο εφαρμογής των συμφωνιών. Μπορεί λοιπόν να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ σημαντικό ρόλο σε έναν πολυμερή διάλογο με την Βόρεια Κορέα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πατσέκο Πάρντο. Τώρα λοιπόν νομίζω ότι ήρθε η στιγμή όπου θα δούμε τι θα γίνει με τους εθνικούς. Είναι η στιγμή δοκιμασίας για αυτούς. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον πρέσβη, τον πρέσβη Χίλ. Με ακούτε? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ακούω. Ε, είμαι στη Φλόριντα και ε, βεβαίως είμαι και εγώ διαθέσιμος για να συζητήσουμε ένα θέμα που το έχουμε συζητήσει επανειλημμένα. Ε, λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά δεν είναι καλή ή δεν ακούμε καλά, οπότε δυστυχώς πρέπει να διακοπεί η διερμηνία. Uh, most importantly, North Korea has a new leadership, Kim Jong-un. I did not believe that the leadership under Kim Jong-il could get any worse. I had not contemplated his son. uh, Ambassador Hill, may I Uh, uh, go in in between for a moment. Colleagues, I'm told by interpreters that there is... The Η πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή. Ε, μου λέγουν οι διερμηνείς ότι δεν είναι σε θέση να ε, μεταφράσουν τα όσα λέτε λόγω και έχεις ποιότητα του ήχου. Δηλαδή μόνο στα αγγλικά μπορεί να γίνει αυτή η ομιλία και δεν θα μεταφραστεί. ώρα. Uh, slowly and I hope uh, people can, uh, can follow me. First of all,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 Δυστυχώς, ε, συγγνώμη που σας είχαμε μόνο σε Skype ε, και δεν μπορέσαμε να κάνουμε τη διερμηνία. Παρ' όλα αυτά χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας ακούσαμε. Ε, συνάδελφοι, έχουμε πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα μπροστά μας, επειδή Έχουμε ένα ακόμη θέμα στην ημερήσια διάταξή μας, πάρα πολύ σημαντικό επίσης. 11.30 ακριβώς πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει με αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Πριν αρχίσει, ε, πριν ανοίξω το λόγο για να θέσετε ερωτήσεις, ε, παρακαλώ σηκώστε τα χέρια σας για να ε, καταρτήσουμε έναν κατάλογο μιλητών, η γραμματεία. Να κάνω κι εγώ εντωμεταξύ την ερώτησή μου το ερώτημά μου είναι προς τον πρέσβη Χιλ όσον αφορά την αξιολόγηση του επίπεδου συνεργασίας μεταξύ Βόρειας Κορέας και Ιράν όσον αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα. Επειδή θα γίνει μια συζήτηση για το JCPOA, αυτή η πληροφορία κατά την άποψή μου είναι σημαντική, πολύ σημαντική, και προς τον δόκτορα Πατσέκο Πάρντο θα ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση. Ποια είναι η άποψή σας σε σχέση με το συνδυασμό αυστηρών κυρώσεων στην Βόρεια Κορέα, απαραίτητο είναι αυτό, με τη δική σας πρόταση εμπλοκής. Πώς θα συνδυαστούν αυτά τα δύο. Και Εγώ έχω τις επιφυλάξεις μου σε σχέση με την συνεργασία στον τομέα του αθλητισμού. Γιατί αν θυμάστε, ε, τα βίντεο και τις φωτογραφίες ε, από την Βόρεια Κορέα, τι να σας πω, είναι μια απλή εκδήλωση της ε, ισχύω της οικογένειας του ηγέτη του Κιμ Ιονγκούν. Οπότε δεν ξέρω, νομίζω ότι αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις δικές μας στρικές πολιτικές. Θα ήθελα να ακούσω λοιπόν τα σχόλιά σας. Christia, you would like to... Κύριε Κριστέ, θέλετε να πάρετε το λόγο τώρα. Λοιπόν, ε, θα έλεγα να ακούσουμε τρεις ε, παρεμβάσεις από τους ε, συναδέλφους και μετά θα ακούσουμε την απάντηση. Πολύ ωραία. Ο κύριος Μποστινάρο. Παρακαλώ κύριε Μποστινάρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω τον πρέσβη κύριο Χίλ να μας πει πώς ακριβώς ε, εξηγεί την ε, τεχνολογική και επιστημονική εξέλιξη της Βόρειας ε, Κορέας, η οποία σε πολύ λίγα χρόνια μπόρεσε να φτάσει σε ιδιαίτερα εντυπωσιακό επίπεδο. Δηλαδή από μια χώρα ε, που είχε πολύ φτωχή τεχνολογία ε, μπόρεσε να φτάσει στο σημείο που έφτασε σήμερα. Τι κρύβεται πίσω από αυτό, γιατί κάποια στιγμή άκουσα από έναν ε, Ρώσο μιλητή ότι στη Βόρεια Κορέα έχουν ένα είδος Silicon Valley για πυρηνικές έρευνες, αλλά χαζομάρες είναι αυτά, εγώ δεν τα πιστεύω. ποιοι είναι εκείνοι που βοήθησαν τη Βόρεια Κορέα να προχωρήσει τόσο γρήγορα. Ο κύριος ε, Ρούμπιχ, έχει το λόγο. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ε, πρέπει να είστε συγγνώμη, καθυστέρησα, γιατί είχαμε ψηφοφορία στην Επιτροπή Ήτρε. Νομίζω όμως ότι είναι πολύ σημαντικό ε, το ότι υπάρχει αυτή η συζήτηση. Και για μένα λοιπόν είναι απόλυτα σαφές ότι θα πρέπει να αναζητήσουμε εναλλακτικές λύσεις. Ίσως αυτό να το πετύχουμε μέσα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και η η άποψή μου είναι πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τον αθλητισμό γενικότερα, να καταστήσουμε δυνατές συναντήσεις, να δημιουργήσουμε ομάδες ενδιαφερομένων οι οποίοι ε, θα συναντιόνται και θα αναζητούν ε, εναλλακτικές λύσεις για να συζητηθούν ε, να χρησιμοποιούμε την πολιτική του καρότου και του μαστιγίου ε, το μαστίγιο φορά τον πρέσβη, αλλά θέλω να ρωτήσω και για τα καρότα. Τι μπορούμε να προσφέρουμε ως καρότο στην Βόρεια Κορέα για να συζητήσει μαζί μας. Έχετε ίσως ένα οπλοστάσιο καρότων που να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Ο κύριος Σαφχάουζε, ε, λυπάμαι που δεν μπορούμε να προσφέρουμε διερμηνία. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι η συζήτηση αυτή περιστρέφεται γύρω από το εξής. Τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα η ΕΕΔ, η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, τι πρωτοβουλία μπορεί να αναλάβει για να μπορέσουμε να ε, προσθέσουμε κάποια αξία. Ποια είναι η ευρωπαϊκή υπεραξία που μπορεί να προσθεθεί εδώ θα πρέπει να δούμε το ιστορικό πλαίσιο καταρχήν. Θυμίζω ότι εμείς είμαστε υπέρ της στήριξης του διεθνούς δικαίου. Και αυτή τη στιγμή μια χώρα δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο, μπαίνουμε σε περιπέτειες. Αυτό το είδαμε ε, και στο Ιράκ και στη Λιβύη και επανειλημμένα και πρόσφατα στην ιστορία μας. Όπου μία χώρα ή περισσότερες, μια συμμαχία κρατών, επεμβαίνουν εκτός διεθνούς δικαίου, στο περιθώριο του δικαίου. Και επειδή η ιστορία επαναλαμβάνεται συχνά αυτή, έχετε χώρες οι οποίες θέλουν οπωσδήποτε να εξασφαλίζουν την ανεξαρτησία τους για να μην εξαρτώνται από μια εξωτερική ε, ισχύ από μια και μόνη χώρα. Και η πυρηνική βόμβα εγγράφεται σε αυτή την ε, επιθυμία ε, ανεξαρτησίας όταν θέλησε η Γαλλία να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, αντιτάχθηκαν οι Αμερικανοί. Επανειλημμένα ε, προσπάθησαν να δολοφονήσουν τον στρατηγό de Gaulle. Γιατί τώρα αυτά είναι δημόσια, ανοίξαν τα αρχεία και ε, χρησιμοποίησαν τον κύριο Μονέ ως Αμερικανό πράκτορα για να μην έχει πυρηνικά ε, η Γαλλία. Μετά Βοηθήσαμε το Ισραήλ να αποκτήσει πυρηνικά, που κατά την άποψή μου είναι καλό πράγμα, αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η ατομική βόμβα είναι ένα στοιχείο ε, κυριαρχίας ε, και μετά το Ιράν, η Βορεια Κορέα που θέλουν να εξασφαλίσουν την ασφάλειά τους και φοβούνται κατά κάποιο τρόπο μήπως τους καταστρέψουν. Αυτά τώρα έχουν βάση, δεν έχουν αυτοί οι φόβοι και άκουσα τον κύριο Πρέσβη πάρα πολύ προσεκτικά είναι γεγονός ότι υπάρχει και μία επιθυμία κατάκτησης, αλλά βασικά φόβος είναι αυτό. Λοιπόν, τι μπορούμε εμείς να κάνουμε αυτή τη στιγμή ως Ευρώπη, το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε ποιο είναι. Ε, κυρίως να μην έχουμε ένα συνασπισμό απέναντι σε έναν άλλον συνασπισμό. Θα πρέπει να πάμε στο Συμβούλιο Ασφαλείας και να μιλήσουμε με την Κίνα, με τη Ρωσία, με τις Ηνωμένε Πολιτείε, με τη Γαλλία, με το Ηνωμένο Βασίλειο και μετά από πρωτοβουλία, γιατί όχι, της κυρίας Μογκερίνη, για να αρχίσει μια συζήτηση γι' αυτό ακριβώς το θέμα. Οι δράσεις, οι κυρώσεις δεν αρκούν, ούτε η εισβολή. Αυτό θα ενισχύσει το καθεστώς στην πυρηνική του πολιτική. Αυτό τα ξέρουμε πολύ καλά. Το δείχνει όλη η ιστορική εξέλιξη με τα καθεστώτα αυτά. Ας αρχίσουμε ένα διάλογο. Αν χρειαστεί αύριο να επέμβουμε δια της βίας, που δεν το αποκλείω, είπε και ο κύριος πρέσβης ότι είναι μια παλιά ιστορία αυτή να θέλει κάποιος να, να κατακτά αυτά που έκανε ο πατέρας του, παππούς του κτλ. Ωραία, τα καταλαβαίνω όλα αυτά, αλλά για να επέμβουμε χρειάζεται μια διεθνή συμμαχία εφόσον έχουμε προετοιμάσει το έδαφος. Και, όχι για ένα νέο παγκόσμιο πόλεμο, αλλά για μια διεθνή συνεννόηση, έτσι ώστε να συγκρατήσουμε και να ανασχέσουμε μια κακόβουλη δύναμη όπως ήταν η Βόρεια Κορέα. Εμείς θα πρέπει να συνεισφέρουμε για να δημιουργηθεί ένας πολυπολικός κόσμος, ε, διάλογος μεγάλων δυνάμεων και όχι να αφήσουμε ε, απέναντι έναν ε, ανεξέλεγκτο παίκτη όπως είναι η Βόρεια Κορέα. Μάλιστα, εδώ ολοκληρώνεται ο κατάλογος των ομιλητών. και θα παρακαλούσα να απαντήσουν οι ε, ομιλητές από το πάνελ με την αντίστροφη σειρά. Πρώτος ο πρέσβης Κρίστοφερ Χίλ και μετά οι υπόλοιποι με την αντίστροφη σειρά από εκείνοι που πήραν το λόγο. Έχετε το λόγο, παρακαλώ, εξοχότατε κύριε πρέσβη.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 made us realize we're not isolated. And in London, we have a community of around 600 North Koreans, the biggest one outside of Asia. And what made them try to escape the country was partly the repression from the regime, but secondly, they saw interaction. Λοιπόν, έχουμε δει εκεί δράσεις και με τους Κινέζους και με τους Ρώσους και με τους Ευρωπαίους. Και νομίζω πραγματικά η οικονομία της αγοράς αναπτύσσεται και στην Πιονιάνγκ. Παλαιότερα ήταν ανέκδοτο αυτό, λέει ο κ. Πατσέκο. Ε, είναι πολύ δύσκολο να ε, κατασταλεί αυτό από το καθεστώς και βασικός λόγος είναι ε, υπάρχει ένα μεγάλο κίνημα ε, απελευθέρωσης της οικονομίας. Έχω ακούσει πολλά και από τους πρόσφυγες και από άλλους. Τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ρωτήσατε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μόνος θεσμός που έχει στρατηγική εταιρική σχέση με την Κορέα, την Ιαπωνία και την Κίνα και διπλωματικές σχέσεις με τη Βόρεια Κορέα. Είναι πραγματικά ο μόνος θεσμός που έχει πρόσβαση στους βασικούς πρωταγωνιστές στην περιοχή εκεί και με τις οικονομίες πολιτικής και η ΕΕΔ και διάφορα θεσμικά όργανα έχουν πραγματικά εμπειρία για τη Βόρεια Ανατολική Ασία. Ε, όσο και αν έχουμε διαφορετική γνώμη εμπειρία, βάσει ο καθένας με τα βιώματά του. Ο, ο δόκτωρ Αντουάν Μποντάς, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Για την πρώτη ερώτησή σας που κάνατε στα γαλλικά, κύριε Σαφαζέρ, για το αποτρεπτικό σκέλος των πυρηνικών και βάσει της ιστορικής εμπειρίας ε, έχει αποτρεπτική ισχύ, συμβατική η Βόρεια Κορέα και ε, ε, μάλιστα είναι μεγάλη διαφορά με τη Λιβύη ε, και με το Ιράκ έχουν όμοιρο ένα εταίρο των Ηνωμένων Πολιτειών είναι πολύ κοντά τους η πόλη της Σεούλ. Ένα από αυτά τα στοιχεία δηλαδή ε, είναι πολύ σημαντικό αλλά και περισσότερο το πολιτικό της νομιμοποίησης ε, του καθεστώτος και ιδιαίτερα του νεαρού ηγέτη γιατί είναι ένα εργαλείο νομιμοποίησης. Συνεχίζω στα αγγλικά. Υπάρχει μια βασική ερώτηση για το ποιε είναι οι επιδιώξεις και οι στόχοι της διεθνούς κοινότητας. Σε μια πρώτη η φάση, η αποπυρηνικοποίηση δεν είναι ρεαλιστικό στόχο. Αλλά, απότερος στόχος ναι, αλλά όχι ε, ο πρώτο. Ο πρώτο είναι το πάγωμα τη ανάπτυξη των δυνατοτήτων, πιο βραχυπρόθεσμη προτεραιότητα κανονικά. Και αυτό είναι δυνατό γιατί δεν αποδυναμώνει ε, την νομιμοποίηση του εσωτερικά του Κιμ. Jong-un και μπορεί να το διαπραγματευτεί. Για την ε, επιθετική χρήση των πυρηνικών όπλων, συμφωνώ με τον πρέσβη. Επίσης θα ήθελα να θυμίσω σε όλους μας ότι το θέμα δεν είναι μόνο στρατιωτικό, είναι και πολιτικό. Και όταν συζητούμε με πάρα πολύ ψηλά ιστάμενους αξιωματούχους, βορειοκορεάτες, ε, κατά κάποιο τρόπο εκείνοι ομολογούν ότι η επανένωση της Κορέας υπό την ηγεσία της Βόρειας Κορέας είναι ο καλύτερος τρόπος να καταστραφεί η χώρα. Δεν μπορεί να απορροφήσει 15 εκατομμύρια νότιο Κορεάτες ο Κιμ Ιονγκ Ουν. 50 εκατομμύρια ε, νότιο Κορεάτες. Δεν μπορούν, να τους ελέγξουν. Ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση ο ρόλος δεν είναι διαμεσολαβητή στο διάλογο, αλλά διευκολυντή να έρθουν πιο κοντά οι χώρες ε, για το διάλογο και με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Μπρέντερ, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Ευχαριστώ πολύ να επιβεβαιώσω ότι από μας, ε, ε, η δική μας προοπτική είναι ότι το βασικό ζήτημα που μας επηρεάζει στο να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε τις χώρες ε, να πάνε σε πυρηνικό πρόγραμμα, μιλούμε για τη Βόρειο Κορέα, μιλούμε και για άλλες χώρες και άλλες καταστάσεις ε, που ε, θεωρούμε ότι θα μπορούσαν να αποτελέσουν επίσης απειλή αν μπορεί να εξελίξει ή να κάνει πράξη την πυρηνική της απειλή η Βόρεια Κορέα. Είναι καθεστώς η Βόρεια Κορέα η οποία ε, εξαρτά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και πώς επιβιώνει με την επιτυχία των πυρηνικών όπλων. Και αυτό είναι δύσκολο γιατί είναι μόνο ζήτημα εξωτερικών υποθέσεων για τη χώρα αυτή. Είναι ένα ζήτημα για το οποίο, με το οποίο έχει συνδέσει την επιβίωση, την, την του το καθεστώς και θα είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό γιατί το κόστος συντήρησης είναι πάρα πολύ ψηλό. Πώς μπορούμε τώρα να επιτύχουμε την αποπυρηνικοποίηση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο υπό το φως όσων ακούσαμε σήμερα είναι πολύ μακριά. Τώρα το πάγωμα τι να σας πω, δεν ξέρω αν είναι εναλλακτική επιλογή. Να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω ε, αν μπορούμε να το εξετάσουμε αυτό το ενδεχόμενο, γιατί υπάρχει περίπτωση, υπάρχει ο κίνδυνος να παραμείνει μόνιμα μετά και ε, είναι ένα νομικό κενό το οποίο δεν θέλουμε να δημιουργηθεί. Και το επόμενο μου ε, σημείο είναι το εξής. Εμείς, εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιβεβαιώσουμε Ένα παίκτη μεταξύ των πολλών. Ε, ενδεχομένως, ε, αν είμαστε σοβαροί για αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα, που ε, ε εμείς δεν είμαστε ο βασικότερος παίκτη, να σας πω την αλήθεια, το να μπορέσουμε λοιπόν εμεί να επηρεάσουμε την πορεία των γεγονότων ε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θέλουμε να συνεργαστούμε με, άλλες, με άλλους για να μπορέσουμε συλλογικά να επηρεάσουμε την πορεία των πραγμάτων. Πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη τι πιστεύουν οι άλλοι και αυτό είναι τμήμα της πολιτικής μας. Η προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που έγκυται. Έχουμε πολλά να προσφέρουμε. Είπαμε, υπόθηκε ότι είμαστε ένα υπόδειγμα του πώς να ε, υπερβεί κανείς μία ε, σύγκρουση. Όντως, πάρα πολλά μαθήματα μπορεί να πάρει κανείς από αυτό και θα μπορούσε να ήταν χρήσιμο σε ένα βαθμό. Αλλά είμαστε σε ένα τμήμα, σε ένα κομμάτι, σε ένα στάδιο της διαδικασίας όπου το μάθημα, αυτό που έχουμε μάθει από όλα αυτά και η ηλική ενίσχυση, η οικονομική συνεργασία που μπορούμε να θέσουμε επιτάφητος. Ε, είναι μεν πολλά και μπορούμε να τα κάνουμε, αλλά πρέπει η σειρά να είναι σωστή. Αν εμπλακούμε, τώρα σε τέτοιες δραστηριότητες, θα νομιμοποιήσουμε το καθεστώς και το πυρηνικό του πρόγραμμα βεβαίως και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θέλουμε να κάνουμε. Οπότε θέλουμε να εστιάσουμε στις κυρώσεις ε, συνεργαζόμενοι παράλληλα με τη διεθνή κοινότητα για να μπορέσουμε η Βόρεια Κορέα τουλάχιστον να αρχίσει κάποια πρώτα βήματα από να υπάρχει ένας αξιόπιστος και ε, ε, πραγματικός διάλογος. Ε, ε, αυτός νομίζω είναι ο καλύτερος τρόπος για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις βασικές μας ανησυχίες να είμαστε σε μεγαλύτερη επαφή με αυτή τη χώρα για να μπορέσουμε μετά να μπούμε σε διαπραγματεύσεις που ενδεχομένως να επιλύσουν το πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Πριν ολοκληρώσω το τμήμα αυτό της συνεδρίασής μας θα ήθελα να πω ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή συζήτηση αυτή που κάναμε, μια συζήτηση ουσίας. Να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και τους προσκεκλημένους ε, εμπειρογνώμονες για τη συμβολή τους ε, σε σχέση με την εξέταση του θέματος θέματος ε, της πυρηνικής απειλής που ε, θέτει πλέον η Βόρεια Κορέα θέλουμε να παρακολουθήσουμε τις διπλωματικές, τη διπλωματική συνέχεια, όπως επίσης και τη συνέχεια των κυρώσεων. Η ακρόαση αυτή είναι πάρα πολύ χρήσιμη στο πλαίσιο της προετοιμασίας ε, των των αποστολών που θα πάνε από την Επιτροπή Εξωτερικών στην Ιαπωνία και στην Νότια Κορέα την επόμενη χρονιά και επειδή είναι η τελευταία μας συνεδρίαση για φέτος θα θέλω να σας ευχηθώ καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος. Ευχαριστώ πολύ. On behalf of uh, subcommittee. Εξ ονόματος της Υποεπιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω ε, όλους τους εξέχοντες ομιλητές μας για τις εξαιρετικές ε, ομιλίες τους καθώς και τους ερμηνείς που προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα με αυτές τις τεχνικές δυσκολίες. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και σας κύριε Πρέσβη που ξενυχτάτε. Παρακαλώ μην φύγετε συνάδελφοι, έχουμε και συνέχεια. Άλλο ένα θέμα και σημαντικό ε, στην Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας για την κλιματική αλλαγή. Ένα πάρα πολύ μικρό διάλειμμα για να αλλάξει το πόντιο του Προεδρείου. Ladies and gentlemen, please be seated. Καθίστε παρακαλώ κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ. Το τελευταίο σημείο λοιπόν στην ημερήσια διάταξη, το τελευταίο ουσιαστικό σημείο της συνεδρίασής μας. Privilege ε, είναι το σημείο υπαριθμών 6. Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας παρουσιάζω ε, το θέμα αντιμετώπιση προκλήσεων νέου τύπου, η κλιματική αλλαγή στην αρκτική περιοχή και οι γεωπολιτικέ συνέπειε των προηγουμένων ενεργειακών τεχνολογιών. Uh, the, geopolitical... Είναι γεωπολιτικό βεβαίως ε, σημαντικό σημείο και έχουμε και προηγμένες ενεργειακές τεχνολογίες. Έχουμε τρεις εξέχοντες ε, ομιλητές ε, που ε, προσωπούν το Στρατιωτικό Συμβουλευτικό Συμβούλιο του Κέντρου Ναυτικών Αναλύσεων των ΗΠΑ. Αντιπρόεδρος ηγείται της αντιπροσωπείας. Ο αντινάβαρχος Λι Γκάν, αντινάβαρχος εν αποστρατεία ε, του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού. Έχουμε τον στρατηγό Donald J. Hoffman, που επειδή είναι στην αεροπορία είναι πτέραρχος και μέλος επίσης ε, του Στρατιωτικού Συμβουλευτικού Συμβουλίου και τελευταίος χωρίς καθόλου είναι λιγότερο σημαντικός είναι ο υπονάβαρχος ένα στρατεία του Βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού Νίλ Μωρισέτη. Ε, Κυρίες και κύριοι, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση θα ήθελα να δώσω μέσω στο λόγο. Ξέρω ότι είναι περιορισμένος ο χρόνος και το θέμα εξαιρετικά σημαντικό και ενδιαφέρον. Right. Uh, Deputy Admiral Floris. Βαρχέ, έχετε το λόγο παρακαλώ. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και χαιρόμαστε για την ευκαιρία που έχουμε να συζητήσουμε με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στην υποεπιτροπή σας. Πριν από 10 χρόνια, το Κέντρο Ναυτικών Ενελίσεων έχει συγκεντρώσει στρατηγούς και αντιναβάρχους τριών και τεσσάρων αστέρων, ένα από στρατεία από όλους τους κλάδους των ενόπλων δυνάμεων και την ακτοφυλακή ε, για να ε, συζητήσουμε θέματα που έχουν να κάνουν με την τότε ε, παρατηρούμενη όλο και μεγαλύτερη κλιματική αλλαγή λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Κατά τη διάρκεια των ετών αυτών, από το 2006 μέχρι το 2007, ε, το Στρατιωτικό Συμβουλευτικό Συμβούλιο, γιατί έτσι αποκλήθηκε αυτό το όργανο, κατέληξε ότι πραγματικά υπήρχε απόλυτη σχέση μεταξύ των κλιματικών αλλαγών και ε, της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ. Από πολλούς ε, σκοπούς και λόγους και για πολλές πτυχές. Παρέμεινε αυτό το συμβουλευτικό όργανο, άλλαξε όμως σύσταση και σύνθεση. Τώρα είμαστε καμιά τριανταριά που έχουμε υπηρετήσει ε, στο CNA, το Στρατιωτικό Συμβουλευτικό Συμβούλιο, στο Κέντρο Ναυτικών Αναλύσεων. Έχουμε κάνει πολλές εκθέσεις για την ενέργεια και για την προηγμένη ε, ενέργεια και ποια είναι η οικονομική και στρατιωτική ωφέλεια. Ε, για το πώς θα ηγηθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη μετάβαση σε μια ενεργειακή οικονομία με προηγμένες ενέργειες. Αυτό είναι το ένα στοιχείο που θα αναλύσουμε σήμερα και το άλλο είναι τα νερά. Βεβαίως το Στρατιωτικό Συμβουλευτικό Συμβούλιο ε, εξετάζει τα θέματα αυτά ε, με βάση την εθνική ασφάλεια και τη στρατιωτική όμως αποτελεσματικότητα. Εκεί δίνεται η έμφαση. Οι προηγμένες τεχνολογίες βεβαίως από τη μία μας ενδιαφέρει να βελτιώσουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο Αμερικανικός στρατός και από την άλλη να εντοπίσουμε τις εξελίξεις εκείνες και τις διπλωματικές οδούς και διάβλους που συνδέονται με την προηγμένη ενέργεια για να μειωθεί η ζήτηση για ε, επιχειρήσεις των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Βεβαίως ανησυχούμε για κάποιες παραδοσιακές απειλές. Τέσσερις οι χώρες είναι κυρίως προκλήσεις. Βόρεια Κορέα, Ρωσία, Ιράν και ενδεχόμενη ε, ανταγωνίστρια ε, αναδυόμενη η Κίνα. Αλλά ανησυχούμε πάρα πολύ για βίες εξτρεμιστικές οργανώσεις. Δηλαδή τέσσερα συν ένα λέει το Πεντάγωνο ότι είναι οι απειλές. Τέσσερα κράτη και το ένα είναι ε, οι μη κρατικέ οντότητε που εμφανίζουν μεταστάσει. Ε, και βλέπουμε ότι συνδέονται αυτά με την τροφή και με το νερό, θέματα εθνικής ασφάλειας, δημογραφικό, ενέργεια, κλιματικές αλλαγές. Όλα αυτά επηρεάζουν τον είδο, το είδος των δυνάμεων που θα πρέπει να έχουμε και να κληθούν να υπηρετήσουν και ε, τις συνθήκες υπό τις οποίες θα επιχειρούν και θα λειτουργούν. Σε μία έκθεση του, διεθνου, του Εθνικού ε, Συμβουλίου Πληροφοριών για τις τάσεις της παγκόσμιας του 2030 προβλέπεται ότι μέχρι τα μέσα του αιώνα, περίπου μέχρι το 2050, η ζήτηση ενέργειας θα αυξηθεί παγκοσμίως κατά 50% και το νερό κατά 40% για τρόφιμα 35%. Όλα αυτά καταδεικνύουν ότι υπάρχουν κάποιοι τομείς ε, που πραγματικά στερούνται πόρων και εκεί θα αυξηθεί η ζήτηση. Γιατί βασικός στόχος, μάλλον βασικός λόγος ε, αυτής της αυξανόμενης ζήτησης είναι η αύξηση του πληθυσμού. Αλλά αυτά όλα δεν είναι γραμμικά. Διότι υπάρχουν προσδοκίες, υπάρχουν επιθυμίες να βελτιώσει κανείς το επίπεδο διαβίωσης και να βρει μια καλύτερη μοίρα και αυτό θα παίξει σημαντικό ε, ρόλο σε αυτές ε, τις τρεις ε, αυξανόμενες ζητήσεις για νερό, ενέργεια και τρόφιμα. Έχουμε λοιπόν μια ε, νέα τεχνολογία προηγμένη και οι ανάγκες ενέργειας προς το παρόν καλύπτονται από τα ρηκτά καύσιμα. Θα δώσω το λόγο στον επόμενο ομιλητή, Πτέρα Αρχέ, για να σας μιλήσει για την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ σήμερα. Η ενέργεια ήταν πάντοτε κρίσιμο στοιχείο της εθνικής ασφάλειας αλλά και της παγκόσμιας ασφάλειας ε, ε, γιατί μπορεί μια στρατιωτική δύναμη να πάει να πολεμήσει ε, για την ενέργεια και δίνει τη δυνατότητα να επιβιώσει στην μάχη και να επιστρέψει κιόλας ε, από τις επιχειρήσεις της. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα και για τις περιφερειακές οικονομίες. Ε, είναι σημαντικό για την ανάπτυξη, ακόμη και για το... Για... Ακόμη, για όλες τις ένοπλες δυνάμεις είναι πάρα πολύ σημαντική η ενέργεια. Εξαρτώμεθα από την ενέργεια. Έχουμε καταναλώσει ενέργεια κυρίως ε, σε υγρή μορφή, χωρίς να σκεφτόμαστε τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Η ενέργεια μας έχει επιτρέψει, να αναπτυχθούμε, να ευημερούμε σε κάποια σημεία ε, του κόσμου, αλλά υπάρχουν βέβαια και κάποια μειονεκτήματα. Πρώτα απ' όλα το περιβαλλοντικό ε, ζήτημα και επίσης ε, πού υπάρχει και πού δεν υπάρχει. Υπήρχε, λοιπόν, υπήρξε λοιπόν χρήση βίας πολλές φορές όταν έλειπε η ενέργεια, το γνωρίζετε και εσείς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αρκετή αρκετή ενέργεια και πολλές φορές και εμεί ε, στι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαμε. Ε, έχουμε λοιπόν μια, ένα παράθυρο ευκαιρία με την υδρορογμάτωση, με το σχιστολιθικό αέριο, με μη συμβατικές ε, με μη, συμβατικές, μη συμβατικούς τρόπους εξόριξης ενέργειας, πράγματα τα οποία είναι δύσκολα να τα αντλήσουμε, μας δίνει μια βεταβατική περίοδο για να περάσουμε σε προηγμένες τεχνολογίες. Εμείς θεωρήσαμε ότι η προηγμένη ενέργεια είναι πιο καθαρή, πιο ε, αποδοτική, ε, όπου τη χρειαζόμαστε, όχι παντού και πρέπει να πω ότι τουλάχιστον από την πλευρά ε, των ενόπλων δυνάμεων ε, είναι αλήθεια ότι και τα πολεμικά πλοία και τα πολεμικά αεροσκάφη θα χρειαστούν υγρή ενέργεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Παρόλα αυτά μπορεί να υπάρχει μια πιο καθαρή ενέργεια που θα έχει παρόλα αυτά ένα περιβαλλοντικό αντίκτυπο για κάποιο χρονικό διάστημα. Ε, μέχρι να, έρθουν, να, έρθει, να έρθει το Star Wars θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για μας να ε, ε, να βρούμε κάποια άλλη λύση. Ε, η βασική πηγή ενέργειας είναι ο ήλιος. Είτε είναι ο ήλιος ηλιακή ενέργεια από μόνη της ή περιμένουμε ο ήλιος να δημιουργήσει αέρα για να έχουμε ολική ενέργεια. Ε, ο ήλιος είναι η βασική μας ε, ε, ενέργεια. Σε κάποιες εφαρμογές μπορεί να υπάρχουν κάποιοι μικροί πυρηνικοί αντιδραστήρες με πάρα πολύ, καλό, πάρα πολύ καλές προδιαγραφές ασφαλείας. Έχουμε επίσης επίγουσες, επίγοντα μάλλον προγράμματα εκτάκτου ανάγκη σε περίπτωση που δεν λειτουργεί κάτι. Δεν ξέρουμε πάντως η τεχνολογία τι θα μα φέρει. Δεν είναι μόνο η πηγή ενέργεια, είναι πώ γίνεται η διανομή τη, πώ την επεξεργάζεται κανεί, πώ την αποθηκεύει. Η αποθήκευση είναι μία από τι βασικότερε αλλαγέ που θα προκύψουν. Ε, η ε, αποθήκευση των μπαταριών, για παράδειγμα. Το βλέπουμε αυτό κάθε μέρα. Ε, και στην Αυστραλία ακόμη είναι ε, μια τεχνολογία που αναπτύσσεται πολύ γρήγορα και εμείς ε, ε, από στρατιωτικής πλευράς θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει μια καλύτερη χρήση ακόμη και στο πεδίο μάχης. Χρησιμοποιούμε λοιπόν αυτό το παράθυρο ευκαιρίας όχι μόνο να καταναλώσουμε την ενέργεια που έχουμε στη χώρα μας αλλά και να τη χρησιμοποιήσουμε μεταβατικά για να είναι πιο αποτελεσματικές οι ένοπλες δυνάμεις και οικονομική μας ε, εξάρτηση από την ενέργεια να είναι μικρότερη, ώστε να υπάρχει μικρότερη πιθανότητα ε, διακοπής της ε, προμήθειας ενέργειας, ώστε η ενέργεια να είναι ένα κομμάτι που θα επηρεάζει λιγότερο ολόκληρη την εξίσωση. Εγώ θα έλεγα ότι η ο εκδημοκρατισμός της ενέργειας είναι πολύ σημαντικός. Ε, δεν μιλάμε για την ενέργεια πια ως πηγή σύγκρουσης ε, ή ε, ιδιοκτησίας. Είναι κάτι το οποίο πρέπει ισότιμα να κατανέμεται. Εν πάση περιπτώσει όχι ισότιμα, αλλά πρέπει να φτάνει η ενέργεια που χρειάζεται, να υπάρχει αρκετό απόθεμα ώστε να μπορούμε να καλύψουμε περιόδους διακοπής προμήθειας ενέργειας. Αυτή ήταν η δική μας μελέτη, αρκετά αισιόδοξη αισιόδοξα είναι τα αποτελέσματα. Βλέπουμε την κατάσταση που ισχύει τώρα. Μπορούμε να είμαστε απεσιόδοξοι βάσει των γεγονότων που βλέπουμε. Δεν μπορέσαμε να προοδεύσουμε όσο θα θέλαμε σε μερικού τομεί. Όμω υπάρχουν ραγδαία αναδυόμενε ευκαιρίε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρο. Ε, και εγώ ευχαριστώ. Θα ήθελα τώρα να κάνω μία παρατήρηση πριν πάμε στον τρίτο μας ομιλητή. Δυστυχώς ε, ε πρέπει να ταξιδεύσω και πρέπει να ταξιδέψω και να φύγω νωρίτερα ε, για να ε, φτάσω στο αεροδρόμιο, πρέπει να πάω στο Βίλνιους, μια πάρα πολύ σημαντική διάσκεψη που αφορά την ασφάλεια. Η κυρία Λέζινγκ, η αντιπρόεδρος, θα, μας, ε, θα με αντικαταστήσει. Μεταδίδεται και στο διαδίκτυο η ακρόαση. Δυστυχώς δεν θα μπορέσω να ακούσω τις απαντήσεις σας, αλλά θα ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση για τις νέες τεχνολογίες που δίνουν κάποια ελπίδα σε σχέση με τον άνθρακα, για παράδειγμα, και τι τεχνολογίε που συμπεριλαμβάνουν άνθρακα, τον καθαρό άνθρακα, εν πάση περιπτώσει. Θα ήθελα να μα πείτε μερικά πράγματα γι' αυτό. Ε, λυπάμαι πάρα πολύ που πρέπει να αποχωρήσω. Θα ήθελα να μείνω μέχρι το τέλος, αλλά δυστυχώς ε, έχω ανηλυμένε υποχρεώσεις. Επόμενος ομιλητής, ε, ε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, υπονάβαρχος Μοριζέτη. Για όσους λοιπόν είχαν την ευκαιρία να δουν ε, κάποιες από τις εκθέσεις, ε, έχουν ε, συσταθεί περίπου 8-9 εκθέσεις, θα εντυπωσιάσει το γεγονός ότι κυρίως όλα αυτά απευθύνονται στις Ηνωμένε Πολιτείες εκθέσεις ε, έχουν ε, κατ' ουσίαν συσταθεί ε, για τις Ηνωμένες Πολιτείες, για την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτείων. Αλλά εγώ θέλω να επισημάνω ότι η τελευταία έκθεση που δημοσιεύτηκε στο Λονδίνο αυτή την εβδομάδα αφορά το θέμα των επιπλοκών που να υπάρξουν από το είδωρ. Αυτό έχει πολύ μεγαλύτερες επιπτώσεις. Ε, εμείς ε, στην Ευρώπη ε, ανησυχούμε πολύ περισσότερο για το θέμα αυτό, πολύ περισσότερο από ό,τι οι Ηνωμένε Πολιτείε. Και θέλω να επισημανώ ότι εδώ υπάρχουν τρεις στρατιωτικές δυνάμεις, όμως το θέμα δεν είναι στρατιωτικό. Είναι ένα θέμα που έχει σχέση με την ασφάλεια ευρύτερα και οι συνέπειες αυτού του θέματος είναι κυρίως οικονομικές και κοινωνικές. οι επιπτώσεις στη ζωή των ανθρώπων από την αλλαγή του κλίματος στο βόρειο και το νότιο η σημερινό. Εκεί υπάρχουν προβλήματα, προβλήματα στη διατροφή, σε πολλά θέματα της καθημερινότητας. Οι επιπτώσεις λοιπόν γίνονται ορατές σε ολόκληρο τον κόσμο. Στην Ευρώπη ε, βλέπουμε την ε, καταστροφή της αλυσίδας ε, διατροφής, την ε, διακύμανση των τιμών των πρώτων υλών, κυρίως της ενέργειας. Βλέπουμε ότι χάνονται αγορές. Πολλές από τις αναδιόμενες αγορές αντιμετωπίζουν πρόβλημα. βλέπετε, ακούμε ότι αυτά τα οποία διαδραματίζονται είναι ε, στο, νερό στο μήλο των ακραίων οργανώσεων. Για μας λοιπόν τίθενται πάρα πολλά ερωτήματα. Το πρώτο εξ αυτών είναι ότι η αλλαγή του κλίματος είναι ένας παράγων που συμβάλλει στην αστάθεια ανά τον κόσμο. Αυτό είναι προφανές. Όμως ε, πρέπει να διουργηθούμε πόσο καλά είναι τα συστήματα της έγκαιρης ε, προειδοποίησης. Ε, προσπαθούμε να δούμε θέματα παραδοσιακά, αλλά πρέπει και να κατανοήσουμε τι συμβαίνει όταν αυξάνονται οι τιμές, όταν οι άνθρωποι μετακινούνται, όταν υπάρχουν προβλήματα λειψιδρίας. Η στρατηγική μας είναι ολοκληρωμένη, γιατί πολύ συχνά ε, αναφερόμαστε σε εθνικές ε, πολιτικές, υπάρχει μια απειλή και πολλοί καλούνται να αντιμετωπίσουν τους απειλές, αλλά αυτό ε, πρέπει να γίνει με ευρύτερο τρόπο, να αντιμετωπιστούν οι παραδοσιακές και οι μη παραδοσιακές απειλές. Επίσης πρέπει να διορτηθούμε κατά πόσον οι απαντήσεις που δίνουμε είναι συλλογικές ή όχι. Έχουμε στρατιωτικές φωνές, αλλά αυτό που ενδιαφέρει είναι ότι ολόκληρη η κοινωνία πρέπει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Να δούμε αν υπάρχουν στοχευμένες απαντήσεις και κατά πόσον είμαστε πρόθυμοι όλα αυτά να τα αντιμετωπίσουμε ως ένα μακροπρόθεσμο θέμα mainstream και να το ε, εξετάσουμε ως τέτοιο. Γιατί σήμερα πολλοί ασχολούνται περισσότερο με τα βραχυπρόθεσμα και όχι τα μακροπρόθεσμα θέματα. Και τέλος ε, πρέπει να διορτηθούμε κατά πόσον υπάρχει ε, λύση ασφάλειας ε, στην κλιματική αλλαγή. Αυτά είχα να πω και σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ θα μιλήσω γερμανικά και όσοι χρειάζονται τη διερμηνία παρακαλώ να φορέσουν τα ακουστικά τους. Δυστυχώς ε, η σημερινή συνεδρίαση είναι θύμα ε, το ότι παράλληλα τρέχουν πολλές άλλες συνεδριάσεις και είμαι η μόνη βουλευτής που παρήσατε και θα κάνω και μία ερώτηση. Η κατάσταση στην Αρκτική είναι το αποτέλεσμα ενός παραδόξου. Από τη μία λοιπόν ε, έχουμε την κλιματική αλλαγή η οποία είναι υπεύθυνη αλλά από την άλλη γίνεται και λόγος ε, για το πώς ακριβώς μπορεί να υπάρξει περαιτέρω χρήση των αποθεμάτων ε, πετρελαίου και αερίου. Κυρίως διότι η περαιτέρω χρήση των ορυκτών καψίμων μπορεί να συνεχιστεί, κάτι το οποίο όμως ε, θα οδηγήσει στο ίδιο αποτέλεσμα. Εγώ προσωπικά πιστεύω και έτσι πιστεύει και η πολιτική μου ομάδα ότι η στόχη μείωση κατά 2% στα προβλήματα του κλίματος, αυτό είναι το ελάχιστο, το απόλυτο ελάχιστο. Βεβαίως και έχουμε λάβει υπόψη μας ε, τις ανησυχίες των ε, αυτόχθονων παρότι από την άλλη πλευρά υπάρχουν και ελπίδες και αυτοί να συμμετάσχουν στην ευημερία. Όμως υπάρχουν και άλλα διαφορετικά συμφέροντα, διαμέτρου αντίθετα, φαύλος κύκλος δηλαδή. Και όταν υπάρχει φαύλος κύκλος ε, τίθεται το ερώτημα κατά πόσον είναι δυνατόν να εξευρεθούν ε, ε, λύσεις για να βγει κανείς από το φαύλο κύκλο. Κατά την άποψή μου το ίδιο ισχύει και για την ε, όλο και μεγαλύτερη στρατιωτικοποίηση αυτές της περιοχής. Αυτές όλες οι εξελίξεις δεν μας χαροποιούν ιδιαίτερα. Νομίζω ε, συμφωνούμε όλοι σε αυτό, στο βαθμό βέβαια που υπάρχει και ανθρώπινος παράγοντας. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να σας ερωτήσω το εξής. Κατά τη δική σας άποψη, Υπάρχει μόνο μία δυνατή εξέλιξη. Να το πω, ε, παραδείγματος χάνει και κάτω από το πρίσμα του αγώνα των εξοπλισμών ή των ε, ανταγωνισμών, πολεμικών ανταγωνισμών σε αυτή την περιοχή. Κλαγκές όπλων ακούγονται και διαρωτώ με, αυτά μπορούν να δεσμεύσουν ε, τις ε, παράκτιες χώρες που έχουν άμεσα ενδιαφέρον στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων και των ε, γηγενών πληθυσμών. Και τι βήματα μπορείτε να σκεφτείτε προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι ώστε να μπορεί κανείς να ακολουθήσει δύο κατευθύνσεις, όχι μόνο μία. Αν δηλαδή δεν μπορούν όλοι να συμφωνήσουν ότι στην περιοχή αυτή πρέπει να αποφευθεί οποιαδήποτε μορφή στρατιωτικοποίησης. Κάτι το οποίο κατά τη δική μου άποψη είναι και η καλύτερη λύση. Σας ευχαριστώ πολύ. Δύσκολο ε, ερώτημα ή μάλλον σύνολο ερωτήσεων για να απαντηθεί. Οι Ηνωμένε Πολιτείε πρόσφατα ολοκλήρωσαν το έτος προεδρίας που τους αναλογούσε στο Συμβούλιο της Ρακτικής και γνωρίζω ότι πολλά από τα θέματα αυτά συζητήθηκαν εκεί. Στη Βόρεια Αμερική υπάρχει και ο Καναδάς, όπου φυσικά έχει μεγάλη κυριαρχία στην περιοχή. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν ενδιαφέρον εκεί και συμφέροντα αλλά είναι προετοίμαστες ουσιαστικά να τα διεκδικήσουν, κυρίως εκεί για το προσεχές μέλλον. Γιατί δεν έχουμε στόλο παγωθραυστικών. Αν ε, χρειαστεί ε, πιο εντατική εκμετάλλευση της ακτικής, εάν υπάρξει πρόσβαση εκεί, τότε χρειάζεται και κάπως να πλαισιώνονται ε, όσοι διέρχονται από την περιοχή, είτε για λόγους εμπορικούς, για εξόριξη, είτε για άλλους. Να υπάρχει μια ε, ασφάλεια τους όταν δραστηριοποιούνται και ακόμα και για τον τουρισμό, που όλο και περισσότερο αυξάνεται. το στρατιωτικό συμβουλευτικό συμβούλιο ακόμα δεν έχει μελετήσει εκτενώς την Αρκτική. Εμείς μιλούμε για την ε, διάνοιξη των διόδων εκεί ως έναν επιπλέον παράγοντα στις αλλαγές που παρατηρούμε στο γεωστρατηγικό τοπίο γενικά, που απορρέει από την κλιματική αλλαγή. Δεν έχουμε όμως ε, μελετήσει πάρα πολύ ε, το μέλλον σε ό,τι αφορά με το τι πρέπει να γίνει. Για τα, κατά την άποψή μου, και είναι προσωπική γνώμη αυτή τώρα, αυτή τη στιγμή ένα είναι το κράτος που στρατιωτικοποιεί, ιδιαίτερα στην Αρκτική, η Ρωσία, που εντείνει μάλιστα τις στρατιωτικές προετοιμασίες εκεί. επισκευάζουν βάσεις στις βόρειες περιοχές και πραγματικά η Ρωσία έχει μια πολύ επεκτατική και επιθετική στάση εκεί. Έχει στόλο πάγο και τα μισά περίπου από τα 12 που έχει είναι και πυρηνοκίνητα. Οπότε Κατά την άποψή μου δεν υπάρχει ακόμα ισχυρισμός η αξίωση ε, ε, για προθέσεις ε, της Ρωσίας να κυριαρχήσουν στη Ακτική. Από την άλλη είναι δύσκολο να μην δει κανεί πώς προετοιμάζονται. Προσωπικά συμμερίζομαι την επιθυμία σας η Ακτική να είναι μια περιοχή χωρίς συγκρούσεις και σειράξεις, αλλά και πάλι προσωπική μου άποψη είναι ότι το κόστος εξόριξης πόρων ενεργειακών, μιλώ για ορυκτά καύσιμα από την Αρκτική, θα είναι αρκετά υψηλό ώστε να μην συμφέρει από τις σημερινές τιμές του πετρελαίου. Ωστόσο υπάρχει ένα παράδειγμα που θα μπορούσε να συνηγορήσει προς τη διαχείριση μιας ε, περιοχής με ακραία καιρικά φαινόμενα και έτσι γίνεται και στην Ανταρκτική που υπάρχει πολύ μεγάλη συνεργασία με πολλά κράτη να εκπροσωπούνται και εξ όσων γνωρίζω μέχρι στιγμής ήταν αμοιβαία υποστηρικτική και χωρίς συγκρούσεις η διαχείριση στην Ανταρκτική. Ο Πτέραρχος, συμφωνώ ότι ο περισσότερος ε, ο κόσμος δεν έχει τη στρατιωτική δυνατότητα να ανταποκριθεί στην Αρκτική. Από την άλλη όμως, μόνο ο στρατός και ένα ένοπλες μπορούν να αναλάβουν αυτές τις προκλήσεις που απορρέουν από την ε, λειτουργία εκεί. Αν χρειάζεται διάσωση κάποιου, πούμε, και παγώσει ε, το νερό πριν μπορέσεις να τον εκενώσεις, ε, με διάφορα προβλήματα υγείας, τραυματισμούς και τα λοιπά. Το αμερικανικό ναυτικό το κοιτάει αυτό από πλευρά στρατιωτικής για το πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε σε τέτοιες περιόδους και περιστάσεις κρίσης. Τι γίνεται ας πούμε όταν υπάρχουν κάποιες ε, εξέδρες άντλησης πετρελαίου στα ανοιχτά της Αλάσκας και υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα σπάσει και πρέπει να εκενωθεί το προσωπικό. Δηλαδή δεν είναι στρατιωτική συζήτηση για τη στρατιωτικοποίηση, αλλά και για τη διάσωση. Η διπλωματία και η πολιτική ε, θα πρέπει να προβλέψουν για την εμπορευματοποίηση της περιοχής που θα γίνει, γιατί όσο φθήνουν οι πόροι ε, θα είναι όλο και πιο ελκυστική η εξόριξη ε, που μπορεί να γίνει με τρόπο συντεταγμένο ή με τρόπο άναρχο που να πηγαίνει ο καθένας και να αρπάζει κάτι από εκεί. εκεί πάντως επιστημονική συνεργασία υπάρχει. Αλλά όταν ε, ε, η συζήτηση γίνεται για τα οικονομικά, δυσκολεύουν τα πράγματα. Πάντως πρέπει να γίνει ε, επαφή σε επίπεδο διπλωματικό και πολιτικό. Δύο σύντομα σχόλια Κύριε κύριος Μωρισέτη, όταν ήμουν ειδικό εντεταλμένος για την κλιματική αλλαγή τη κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου και πήγα να συζητήσω το θέμα της Αρκτική. ήταν πολλές οι απόψεις γιατί θα γίνει στο μακρινό βορρά, ε, άμεσα, πιο μακροπρόθεσμα, αργότερα, ποια θα είναι η εντατική χρήση ή όχι. Ε, αν θα γίνει με τρόπο εύσχημο και καλόβουλο ή αν θα υπάρξουν σειράξει. Αυτό που ε, ήταν κοινή αντίληψη ήταν ότι πρέπει να γίνει μια διακυβέρνηση με τρόπο συντεταγμένο ε, και ελεγχόμενο για να μπορέσουμε να ξορίξουμε και ορυκτούς πόρους κτλ. Σε ό,τι αφορά εκεί τα ορυκτά καύσιμα συμφωνώ με τον Ναυαρχό. Το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να μην τα εξορίξουμε καθόλου να δούμε τι γίνεται με την ε, ανανεώσιμε αλλού, με την αποθήκευση, έτσι ώστε να μην είναι ε, οικονομικά σκόπιμο, λογικό, να τρέχουμε εκεί να βγάζουμε ε, πετρέλαιο και φυσικό αέριο από την Αρκτική. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Λούζινγκ. Σίγουρα θα είχαμε πολλά να πούμε ακόμα, πολλά σημαντικά σημεία για μελλοντική συζήτηση. Θα ήθελα να κάνω μια συμπληρωματική ερώτηση. Για τη μελέτη που ανέφερε ο Πτέραρχος, πότε μπορούμε να, να υπολογίζουμε για τη μελέτη, τη μελέτη αυτή να έρθει. Όχι ο Πτέραρχος, συγγνώμη, ο Αντινάβαρχος Λίγκαν. Έχετε πληροφορίες για το ποιος συμμετείχε σε μια τέτοια μελέτη, ποιος ε, έπρεπε να συμμετέχει σε μια τέτοια μελέτη και οι προοπτικές αυτές της διακυβέρνησης της Αρκτικής θα περιλάμβαναν και άλλα στοιχεία. Όχι μόνο στρατιωτικά, οικονομικά και οικολογικά, αλλά θα ήταν και ε, κοινωνιολόγοι, πολιτικοί, επιστήμονες. Ποιοι συμμετέχουν σε μια τέτοια μελέτης. Uh, το Στρατιωτικό Συμβουλευτικό Συμβούλιο θα ε, εξετάσει βεβαίως και επιπλέον ζητήματα σε σχέση με τον αρκτικό κύκλο. Ε, το Εθνικό, Συμβούλιο, το Εθνικό Ερευνητικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Πολιτειών είτε το έχει ήδη κάνει είτε θα το κάνει, μία επιπλέον μελέτη ε, θα εκπονήσει σε σχέση με τις προοπτικές των ΗΠΑ αλλά και τις ε, ε, κοινωνικές, οικονομικές και γεωπολιτικές πτυχές του αρκτικού κύκλου. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να δεσμευθώ εκ μέρους του Κέντρου Ναυτικών Αναλύσεων, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα γίνει σωστά. Έχουμε αναφέρει ότι το βασικό κίνητρο για την εκπόνηση μελετών του Στρατιωτικού Συμβουλευτικού Συμβουλίου είναι η κατανόηση των συνεπειών του μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος μας και επίσης ε, η υποβολή συστάσεων ε, ε, αλλαγών ε, που θα καταστήσουν ε, το στρατιωτικό τομέα πιο αποτελεσματικό. Παράλληλα όμως κάνουμε σχόλια και για κοινωνιοοικονομικά ζητήματα σε ολόκληρο τον κόσμο. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό, αλλά νομίζω ότι θα τα αφήσουμε στους επιστήμονες σε εθνικό επίπεδο να μας δώσουν τα μέσα μέσω της εκπόνησης ε, μελέτης για να ορίσουμε τις, ε, ε, τις συνέπειες για την εθνική ασφάλεια. Ίσως για μας, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, να υπάρχει δυνατότητα να συμβάλλουμε και εμείς σε αυτή τη συζήτηση. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να κλείσουμε τη συνεδρίαση, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά ε, όλους σας και θα ήθελα να κλείσω, όπως σας είπα, τη συνεδρίαση ανακοινώνοντάς σας ε, την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο μια έκτακτη συνεδρίαση της ε, Επιτροπής ΣΕΝΤΕ την Τρίτη λοιπόν 9 το πρωί με 10 θα έχουμε αυτή την έκτακτη Συγγνώμη, πέμπτη διορθώνει τώρα η πρόεδρος, την πέμπτη θα είναι αυτή η έκτακτη συνεδρίαση. Δεν ξέρω αν έχει ήδη επιλεγεί κάποιο θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λύεται η συνεδρίαση. Γεια σας.